Παρακαλώ, καθίστε. Καλώ Καλώς ορίσατε όλοι. Ξεκινάμε τη συνεδρία της Επιτροπής ζητώντας συγγνώμη για αυτή την καθυστέρηση που οφείλεται στην καθυστέρηση του ε, άτυπου τριμερούς διαλόγου με την Κυπριακή Προεδρία και τον Επίτροπο Τσόλος που έλαβε χώρα στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο και έτσι χάσαμε λίγο χρόνο. Στο μεταξύ θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, στους φίλους μας από την Ένωση Νέων Αγροτών της Λομβαρδίας και από την Ένωση Πικάσο. Καλώς ορίσατε και ευχαριστούμε για την παρουσία σας και τώρα. Επειδή έχουμε και περιορισμένο χρόνο, εφόσον συμφωνείτε, θα ασχοληθούμε και με τους τέσσερις φακέλους μαζί. Τα σημεία λοιπόν 9, 10, 11 και 12 θα τα εξετάσουμε μαζί. Ξέρετε ότι μιλάμε εδώ για την προσχώρηση της Κροατίας, για την ένταξη της Κροατίας, ε, την ενσωμάτωση της στα κείμενα αυτά και δίνω το λόγο στον κύριο Κάπουλα για τους δύο φακέλους ε, ενίες ενισχύσεις και αγροτική ανάπτυξη και μετά στον συνάδελφο για τα άλλα δύο θέματα και βλέπω ότι είναι παρόντες εδώ όλοι οι γενικοί διευθύντες γεωργίας. Αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Χαιρετίζω λοιπόν και τον ε, Διευθυντή κύριο Πρέβε. Αν συμφωνείτε θα μιλήσουμε έτσι Καπούλας, Μισελάντε, Τζοβάνι Λαβία και μετά η Κομισιόν ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να διεκπαιρώσουμε τα θέματα γρήγορα. Εάν το ζητήσουν φυσικά οι συγητέ, ε, θα μπορέσουν να μας ενημερώσουν για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων με τους κοιόδη συγγητές. Συμφωνείτε όλοι, θα προχωρήσουμε έτσι Ξεκινάω δίνοντας το λόγο στον Λουίς Κάπουλα Σάντος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι συνοπτικός, γιατί κατά τη γνώμη μου χρήσιμο θα ήταν να ακούσουμε και τους κοιόδης ηγητές, μια και το έργο είναι κοινό. Και καλό θα ήταν ε, οι συνάδελφοι να συμπληρώσουν οποιασδήποτε παραλήψεις. Θα ξεκινήσω από τον κανονισμό για την αγροτική ανάπτυξη, ανάπτυξη πέθρου. Έχουμε προχωρήσει αρκετά, είχαμε αρκετές συσκέψεις και θα ήθελα να υπογραμμίσω και δεν κουράζομαι να το κάνω το επικοδομητικό πνεύμα που επικράτησε σε όλες αυτές τις συναντήσεις μας. Χάρη σε αυτό το πνεύμα συνεργασίας καταφέραμε να σημειώσουμε αρκετή πρόοδο παρόλο που δεν καταλήξαμε ακόμη σε ε, αποκρισταλωμένες συμβαστικές ε, θέσεις. Καταρχήν, για το θέμα των ε, νέων γεωργών. Μάλιστα, έχουμε μια αντιπροσωπεία, τελική αντιπροσωπεία νέων γεωργών που θα ενδιαφερθεί ιδιαίτερα για το θέμα αυτό. Το θέμα των νέων γεωργών είναι ένα θέμα για το οποίο ουσιαστικά έχουμε καταλήξει σε συμβαστική πρόταση θα έχουμε ενισχύσεις από το, δεύτερο, από το πρώτο και δεύτερο πυλώνα για τους ε, νέους γεωργού. Στον πρώτο πυλώνα θα είναι υποχρεωτικές αυτές οι ενισχύσεις. Θα έχουμε προσάυξη κατά 25% των άμεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο. Και η συμβαστική πρόταση ε, λέει η, ε, προσάυξη αυτή να ισχύει για τα 100 πρώτα εκτάρια των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Σε όλα τα κράτη-μέλη, λοιπόν, αν τελικά συμφωνήσουμε την πρότασή μας το Συμβούλιο και η Επιτροπή, ε, τα πρώτα 100 εκτάρια, ε, τα πρώτα 100 θα έχουν ένα το top-up. Επίσης έχουμε 12% του προϋπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων που θα κρατηθεί για τους νέους γεωργούς και επίσης αποφασίσαμε το μη χρησιμοποιηθέν ποσό από αυτό το 12% από τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιηθεί για τους νέους γεωργούς για να έχουν τα ίδια πλεονεκτήματα οι νέοι γεωργοί, παρόλο που δεν είναι νέοι κατά ανάγκη και στην ηλικία. Σε ό,τι αφορά τους μικροκαλλιεργητές, υπάρχει ευρία συνένεση για το θέμα των μικροκαλλιεργητών. Επίσης προτείνουμε οι μικροκαλλιεργητές που λαμβάνουν λιγότερο από, τα, από 1.500 ευρώ να περιλαμβάνονται αυτόματα στο σύστημα των μικροκαλλιεργητών. Αυτοί βέβαια που δεν θέλουν να, συμπεριληφθούν μπορούν να ζητήσουν να παραμείνουν στο ισχύον σύστημα. Σημαντική πρόοδο σημειώσαμε και στο θέμα της ελαστικότητας μεταξύ των πυλώνων. Και υπάρχει μια προκαταρκτική συμβαστική πρόταση, ώστε να έχουμε μεταφορά ε, μέχρι το 15% των ποσών από τον πρώτο στο δεύτερο πυλώνα. Δεν έχουμε ακόμη συμφωνία για τις ε, μεταφορές του δεύτερου πυλώνα. Οι προτάσεις κυμαίνονται από 5% σε 10%. Σε ό,τι αφορά τώρα τις πληρωμές, τις συνδεδεμένες πληρωμές, ε, φαντάζομαι ότι η τελική συμβαστική λύση ε, θα μείνει κοντά στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προτείνει σύνδεση μέχρι 5% των εθνικών ποσών που για ορισμένες χώρες μπορεί να είναι πάνω από 5%. Ίσως ε, καταφέρουμε να συμβιβαστούμε γύρω από αυτές τις ε, τιμές και τις προτάσεις. Αλλά για τα πιο περίπλοκα θέματα, το θέμα του, το θέμα του κάπινγκ των ανώτατων ορίων είναι πιο περίπλοκο, θα είναι πιο δύσκολη η επιτεύξη συμφωνίας. Συνεχίζουμε βέβαια τις εργασίες, αλλά δυστυχώς υπάρχει τεράστια διάσταση απόψε για το θέμα αυτό. Άλλο περίπλοκο θέμα με διάσταση απόψεων ε, είναι το θέμα του κέπινγκ. Είναι δύσκολο αυτό το θέμα, αλλά τελικά καλύψαμε κάποιες διαφορές και πριν από λίγο ε, ακούσαμε και τη θέση του Συμβουλίου. Πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια συμβεστική πρόταση για το greening, για το πρασίνισμα, να εξασφαλίσουμε ένα πράσινο οικολογικό χαρακτήρα στον πρώτο πυλώνα, πιο απλό όμω και πολύ λιγότερο γραφειοκρατικό για του γεωργού, που να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικέ συνθήκες, να έχει μια ευρωπαϊκή διάσταση και προσέγγιση, αλλά να προβλέπει μια ελαστικότητα και μια διακριτική ευχαίρεια στα κράτη-μέλη, χάρη στην εισαγωγή του συστήματο των ισοδυναμιών. Αυτά προς το παρόν. Τώρα συζητούμε το θέμα της εσωτερικής σύγκλησης. Για το κατά πόσο θα πρέπει ε, να έχουμε σύγκληση ε, των πληρωμών ε, εντός μιας περιοχής, εντός κράτους μέχρι το 2019. Δεν ξέρω αν θα γίνει θα καταστεί κάτι τέτοιο δυνατό. Θα πρέπει πάντως να βρούμε ένα μηχανισμό που θα αποφεύγει στρέβλωση ανταγωνισμού και ταυτόχρονα θα εξυπηρετεί τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά το greening και πάλι, το θέμα της διαφοροποίησης, όπως προτείνεται, δίνει μια κατά τη γνώμη μου ικανοποιητική λύση. Δηλαδή, ε, οι γεωργικέ εκμεταλλεύσεις που έχουν αρδεύσιμη έκταση μέχρι 10 εκτάρια δεν θα υποχρεώνται να ε, εφαρμόσουν το greening. Μεταξύ 10 και 30 εκταρίων αρδεύσιμη ε, καλλιέργεια θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον δύο καλλιέργειες και πάνω από 30 εκτάρια υποχρεούνται να έχουν τρει καλλιέργειες. Τώρα το θέμα της βοσκονομής, έχει, της χορτονομής έχει διευρυθεί, οπότε μια προσωπική χορτονομή μπορεί να είναι ισοδύναμη με καλλιέργεια. Οπότε μπορεί να ενταχθεί στο σύστημα της διαφοροποίησης και η προσωρινή βοσκονομή ως μη επιπλέον καλλιέργεια. Σε ό,τι αφορά τις ζώνες οικολογικού ενδιαφέροντος, ένα άλλο ευαίσθητο ζήτημα. Η πρόταση ε, που βρίσκεται επιτάπητος και εξετάζεται ε, φτάνει μέχρι τα 10 εκτάρια αρδεύσιμης ε, επιφάνειας. Δεν μιλώ για το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης, γιατί είναι αρδεύσιμη μόνο έκταση. Εξαιρούνται λοιπόν από την εφαρμογή αυτού του ποσοστού της ζώνης οικολογικού ενδιαφέροντος, ενώ οι εκμεταλλεύσεις που έχουν πάνω από 10 εκτάρια αρδεύσιμη έκταση. Αλλά αυτή η έκταση είναι πάνω από 20% του συνόλου της αρδεύσιμης καλλιέργειας, της αρδεύσιμης επιφάνειας, τότε θα πρέπει να τηρηθούν οι ζώνες οικολογικού ενδιαφέροντος, μια και δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία επί του συγκεκριμένου ποσοστού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει 7%, ε, άλλε τροπολογίε ζητούν 3%, μερικοί υποστηρίζουν 5%, η Επιτροπή Περιβάλλοντος 7%. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να βρούμε κάποια ισορροπία μεταξύ του 3% και του 7%. Ίσως 5% θα ήταν μια χρυσή τομή. Αλλά μερικές πολιτικές ομάδες, ακόμη και με το 5% έχουν πρόβλημα γιατί θέλω λιγότερο. Ενώ άλλες χώρες, άλλες ομάδες θέλουν περισσότερο, οπότε και αυτές έχουν πρόβλημα. Μπορούμε εναλλακτικά να ψηφίσουμε αυτά τα ποσοστά. Δεν είναι αναγκαίο να συμπεριλάβουμε στη συμβαστική λύση και συγκεκριμένο ποσοστό. Θα μπορούσαμε αυτό να το αφήσουμε κατά μέρο. Αυτά ακροθυγώ αυτή είναι η κατάσταση για τι άμεσε ενισχύσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κανονισμό για την ανάπτυξη της υπαίθρου, την αγροτική ανάπτυξη. Εκεί είχαμε λιγότερα επίμαχα θέματα, ήταν πιο εύκολη η επίτευξη πρόοδου και για πολλά λεπτομεριακά θέματα καταλήξαμε σε συμβαστικές προτάσεις. Εκκρεμούν κάποια προβλήματα βέβαια. Πάντως πιο σημαντικά θέματα όπως η συγχρηματοδότηση των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων που θα είναι 55% η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε 50%. Υπήρχε μία πρόταση για συγχρηματοδότηση 60%. Τελικά η συμβαστική λύση βρίσκεται κάπου στη μέση και πιστεύω ότι θα συμφωνήσουμε με το 55% της χρηματοδότησης. Επίσης θα έχουμε τη δυνατότητα μιας συμβαστικής πρότασης για να απαιτήσουμε 25% του εθνικού ποσού για την αγροτική ανάπτυξη να αφιερωθεί σε άγρο περιβαλλοντικά μέτρα και στην οικολογική γεωργία. Ένα ποσό που είναι λίγο ανώτερο από τα, από τα σημερινά ποσά. Σήμερα έχουμε κατά μέσο όρο 24% για τα μέτρα αυτά. Μια και όμως μιλούμε για μέσο όρο, δηλαδή υπάρχουν κράτη που αφιερώνουν λιγότερο από το 24% του προϋπολογισμού στα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα. Αυτό που προτείνουμε είναι σε όλα τα κράτη-μέλη παραγκλήτως τουλάχιστον 25% του προϋπολογισμού να αφιερωθεί σε αγροπεριβαλλοντικά μέτρα. Υπάρχει συμφωνία για τις ε, ενισχύσεις για τους νέους γεωργούς. Υπενθυμίσαμε ότι η διαπραγματευτική εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό ε, και η βάση για αυτή θα είναι ο ισχύων προϋπολογισμός αλλά υπάρχουν κάποια εκρεμή θέματα για δύο θεμελιώδη ζητήματα. Το θέμα των ζωνών ε, με ε, στοιχεία με για φυσικούς όρους. Υπάρχει διαφορετική πρόταση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φαίνεται ότι και το Συμβούλιο έχει διαφορετική γνώμη. Μόλις πληροφορηθήκαμε ότι το Συμβούλιο και το θέμα αυτό είναι μάλλον ε, πιο κοντά στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ το Κοινοβούλιο διαφωνεί. Η πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά παράταση της ισχύουσας κατάστασης. Κάτι που είναι καθιστά δύσκολη την επιτέξη συμφωνίας. Ένα άλλο εκρεμές θέμα αφορά τη διαχείριση των κινδύνων. Στην Επιτροπή μας η πλειοψηφία είναι υπέρ της διατήρηση του συστήματος αυτού στο δεύτερο πυλώνα, όπω προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια, η Επιτροπή περιβάλλοντο ε, υπερψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία η πιθανότητα μεταφοράς στον πρώτο πυλώνα αυτού του συστήματος της διαχείρισης κινδύνων. Υπάρχουν ε, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και στις δύο λύσεις, αλλά υπάρχει διάσταση απόψε μεταξύ των δύο επιτροπών, Γεωργίας και περιβάλλοντο Και διαφωνία και με το Συμβούλιο, γιατί και στο Συμβούλιο υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία υπέρ της διατήρησης ε, του συστήματος διαχείριση των κινδύνων στο δεύτερο πυλώνα. Σε ό,τι αφορά πάλι αυτό το θέμα, ε, άλλο επίμαχο ζήτημα είναι το θέμα των γεωργικών ασφαλίσεων. Κάποιες πολιτικές ομάδες θέλουν να διαγραφεί του, αποκλεισμό μάλλον, εξαίρεση του θέματο των γεωργικών αποκλήσεων. Άλλοι βουλευτές θέλουν να παραμείνει ε, εντός. Θέλουμε να βρούμε μια συμβαστική λύση, αλλά δεν νομίζω η συμβαστική λύση να απέχει πολύ από την ε, πρώτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συγκεντρώνει πλειοψηφία και στο Συμβούλιο, όπως μάθαμε πριν από λίγο. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτές ε, ήταν σε αδρές γραμμές οι βασικές μας συμβαστικές προτάσεις. Θα ήθελα να εκφράσω τη μεγάλη μου ικανοποίηση για τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών και για το ιδιαίτερα επικοδομητικό πνεύμα και το πνεύμα συνεργασίας που έδειξαν χωρίς καμία εξαίρεση οι σκιώδεις ηγητές, χάρη στο οποίο καταφέραμε να σημειώσουμε πρόοδο. Και είμαι πεπισμένος ότι μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, που είναι η νέα μας προθεσμία για την αποστολή των συμβαστικών τροπολογιών ε, στη μετάφραση, πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να αποκρισταλώσουμε αυτές τις συμβαστικέ προτάσεις και μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου θα έχουμε ε, τις ε, συμβαστικές ε, προτάσεις έτοιμες για μετάφραση. Θα ήθελα επίσης να απευθύνω έκκληση προς όλους τους συναδέλφους είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και καλό θα ήταν να, ε, να συσπηρωθούμε ώστε να διαμορφωθεί μια ευρεία πλειοψηφία στην Επιτροπή μας για τα πιο σημαντικά θέματα. Αν έχουμε μια τέτοια δυνατή πλειοψηφία θα μπορέσουμε τον Ιανουάριο που θα ψηφίσουμε να ξεκινήσουμε ήδη τον άτυπο τριμερή διάλογο με το Συμβούλιο. Μια και η εντολή που θα λάβουμε στην Ολομέλεια του Στρασβούργου ε, θα έρθει το Μάρτιο. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει τις διαπραγματεύσεις έστω και ατύπως να τις ε, ξεκινήσουμε σε προηγούμενο στάδιο ώστε να ολοκληρωθούν όλα αυτά στο πρώτο εξάμεινο του 2013. Θα είναι σίγουρα και για τους... Ευχαριστούμε. Εγώ θα συνέχιζα με το ίδιο σύστημα, δίνω τώρα το λόγο στον Μισελ μετά τον Τζοβανίλαβια και στη συνέχεια θα δούμε ποιοι θα ήθελαν να μιλήσουν. Ελπίζω να αναφερθούν όσοι μιλήσουν και στους τέσσερις φακέλους ώστε να δώσουμε μετά τη δυνατότητα στην Κομισιόν να παρέμβει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως και ο Λουίς θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την ομάδα των σκιωδών και των συνεργατών διότι ακόμη και εάν συμφωνούμε αντιλαμβάνουμε ότι υπάρχει ένα θετικό πνεύμα που επιτρέπει να προχωρήσουμε. Όπως ελέγχθη εχθές από τον George Lyon το θέμα αυτό είναι λεπτό και υπάρχουν πολλώσεις οπότε θα είναι δύσκολο να υπάρξουν ε, συμβιβαστικές προτάσεις που να, ε, στις οποίες να συμφωνήσουν όλες οι πολιτικές ομάδες. Έχω υποβάλει 10 ε, συμβιβαστικές προτάσεις για τα 100 πρώτα άρθρα και εφόσον ε, δεν υπάρχουν ε, όλα συμφωνημένα, δεν συμφωνείται κανένα, αλλά έχουμε δύο θετικά σημεία για τη γεωργία και το, τη διανομή γάλατος στα σχολεία. Ε, υπάρχει ένα πρόβλημα με την με τις προδιαγραφές της αγοράς ε, και τις τιμές αναφοράς και όσον αφορά την δημόσια παρέμβαση. Είναι αρκετά πλήρης ο συμβιβασμός που αναφέρεται σε διάφορα προϊόντα αλλά όλες οι πολιτικές ομάδες δεν έχουν συμφωνήσει σε αυτό το συμβιβασμό. Για την ιδιωτική αποθήκευση επίσης δεν συμφωνούν στο συμβιβασμό όλες οι πολιτικές ομάδες. Θέλω όμως να πω ότι αυτός ο συμβιβασμός δεν καλύπτει έναν κατάλογο προϊόντων διότι είναι πολύ μακρύς ο κατάλογος αυτός και ως εκ τούτου είναι αδύνατο να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία στην λίστα αυτή. Οπότε θα έχουμε χωριστές ψηφοφορίες για κάθε ε, ένα από τα προϊόντα σε αυτόν τον κατάλογο και θα δούμε πού θα υπάρξει μία πλειοψηφία. Υπάρχει μία επιφύλαξη ε, εξετάσεως σχετικά με το ελαιόλαδο και τα οποροκυπευτικά. Συμφωνούμε για το πνεύμα του συμβιβασμού, αλλά ε, όσο δεν έχουμε ε, όλες, όλα τα στοιχεία συμπεφωνημένα δεν μπορούμε να ακυρώσουμε αυτό τον συμβιβασμό. Και τέλος, σχετικά με το κρασί, υπάρχει ε, επίσης ένα συμβιβασμός ευρύς ε, για ε, τις οργανώσεις εμπορίας και αγοράς του κρασιού και επ' αυτού βλέπουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτά είχα να σας πω, αλλά μετά από τρεις συνεδριάσεις των σκιωδών εισηγητών δεν υπάρχουν εκπλήξεις, δηλαδή ε, αυτά τα οποία ελέγχθηκαν ή στην ε, αίθουσα ε, επαναλαμβάνονται και αντικατοπτρίζονται και στις συμβαστικές προτάσεις. Ευχαριστούμε Μισελ. Συνεχίζουμε με τον Τζοβάνι Λαβία. Στο μεταξύ καταγράφουμε τις αιτήσει επεμβάσεων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όσον αφορά τον κανονισμό για τη χρηματοδότηση της κοινή γεωργικής πολιτικής, τον οριζόντιο κανονισμό, πρέπει να πω ότι και σε αυτή την περίπτωση ήταν άριστη η συνεργασία με τους κοιόδης εισηγητές για την επιτευξή συμβιβασμού σε διάφορες τροπολογίες. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων όλες οι ομάδες ε, συμφωνούν με τις συμβιβαστικές τροπολογίες που προτάθηκαν για το πρώτο μέρος. Έχουμε φτάσει μέχρι το άρθρο 56. Όσον αφορά αυτά, δηλαδή του όργανα πιστοποίησης, είτε ο εύρος των προτάσεων, είτε την παρακολούθηση, είτε αφορούν την καινοτόμο τοπική συνεργασία, είτε την στήριξη των επιχειρήσεων και των εκμεταλλεύσεων πιστεύω ότι υπάρχει, υπάρχουν μεταξύ ομάδων κοινέ γραμμές που μπορούμε να επισημάνουμε στην Επιτροπή. Συνεχίζουμε τις εργασίες μας σε σχέση με το θέμα της αιρεσιμότητας όπου εμφανίζονται πιο ακαθόδη ζητήματα όσον αφορά την εφαρμογή της αιρεσιμότητας, της οδηγίας για τα ύδατα και της οδηγίας για τα φυτοφάρμακα. Αλλά πιστεύω ότι και σε αυτά τα θέματα, με τις συνεδρίες των επόμενων ημερών με τους κοιόδες, θα καταφέρουμε να επιτύχουμε αποδεκτές συμβιβαστικές τροπολογίες για όλες τις ομάδες. Ένα ξεχωριστό στοιχείο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι εκείνο που σχετίζεται με την ολοκληρωμένη πρόταση της Κομισιόν για τη διαφάνεια. Όσον αφορά αυτή την πρόταση, σε σχέση με το κείμενο που προτείνει η Κομισιόν, φαίνεται να υπάρχουν δικογνωμίες. Εγώ καταρχάς ήδη με τις τροπολογίες που υπέβαλα υπέδειξα ότι χρειάζεται τροποποίηση της πρότασης της Κομισιόν ώστε να αναδειχθεί το δικαίωμα της προστασίας του ιδιωτικού απορρίτου στην πρόταση της Κομισιόν, διότι θεωρώ ότι δεν είναι σωστό για όλους τους γεωργούς κάθε φορά που λαμβάνουν ένα πόρο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δημοσιεύουν στον ιστότοπο το ποσό και το όνομα και το επώνυμα ενώ για όλους τους άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση. Εκεί λοιπόν θα είχαμε διακριτική μεταχείριση αρνητικά προς τους γεωργούς. Γι' αυτό το λόγο προτείναμε να αντικατασταθεί το όνομα και επώνυμα με έναν κωδικό ο οποίος θα αναφέρεται συγκεκριμένα στο άτομο που εποφελήθηκε από το κονδύλο της κοινής γεωρικής πολιτικής και έτσι θα είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί και το θέμα της διαφάνειας. Και αυτό προσφέρει μια ισορροπία μεταξύ της προστασίας του ιδιωτικού απορρίτου και της ανάγκης για διαφάνεια. Ωραία, ευχαριστούμε Τζοβάνι. Ξεκινάμε τώρα με τις αιτήσει ε, για ομιλία ο Άγνιου, Τέσσε, Σεγκρέσκε και um, Ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήσεις. Ε, προς τον κύριο Καπουλά Ευχαριστούμε για τις προσπάθειές σας ε, που προσπαθείτε να αποκτήσουν κάποιο περισσότερο νόημα αυτά τα ζητήματα του πρασινίσματος ε, στο πλαίσιο των τιμών που έχουμε σήμερα μας ζητούν να καλλιεργούμε με λιγότερο εντατικό τρόπο. Είπατε και θα ήθελα να μου το διευκρινίσετε, είπατε ότι τα πρώτα 10 εκτάρια θα απαλλάσσονται από οικολογικά εστιασμένες περιοχές. Μιλάμε για τα 10 πρώτα εκτάρια οποιασδήποτε εκμετάλλευσης, είτε πρόκειται για νέο αγρότη, είτε για ε, πεπειραμένο αγρότη. Αυτή είναι η πρότασή σα ή αυτά τα 10 εκτάρια χαρακτηρίζονται έτσι ούτω ή άλλως. Και μια γρήγορη ερώτηση προ τον κύριο Λαβία. Είπατε θα υπάρχει ένα κωδικό αντί για όνομα όσον αφορά του παραλήπτες τη ενιαίας ενίσχυση. Ποιο θα έχει πρόσβαση σε αυτόν τον κωδικό. Θα με ενδιαφέρει να μάθω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Άγνιο. Άλμπερντ και Σικέρσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς δεν μπορούσα να παραστώ από την αρχή και άκουσα μόνο τις τελευταίες παρατηρήσεις του κυρίου Κάπολ Σάντο σχετικά με την ρύθμιση αυτή. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που συνέβαλαν σε αυτή την εργασία και ελπίζω να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς που θα επιτύχουν μεγάλες ε, πλειοψηφίες στην Ολομέλεια. Αλλά με το 7% δεν καταλαβαίνω καν την ε, βάση της προτάσεως ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι ξεκινάμε από το τέλος προς την αρχή. Ε, υπάρχει ε, μία ε, υπάρχει ανάγκη ενεργείας, έχουμε υψηλές τιμές ενοικιάσεως γης και θεωρώ ότι όλες αυτές οι προτάσεις είναι αρνητικές. Πρέπει να βρούμε επικοδομητικές προτάσεις και να δούμε εάν το 3, 5 ή 7% θα μπορέσουν να υπερισχύσουν. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι υλοποιήσιμες οι προτάσεις αυτές και το, οι εκτάσεις οι οποίες απαιτούνται και θα πρέπει να ενοικιαστούν ήδη δημιουργούν μεγάλα προβλήματα και από ό,τι διάβασα στο διαδίκτυο ένας ε, ένας γεωργός πρότεινε το χειρότερο, τη χειρότερη γεωργική του ε, έκταση με τη μικρότερη απόδοση για το 7% ε, και κουνάω και εγώ το κεφάλι μου. Θα ήταν πολύ καλύτερο να μπορεί κανείς να κάνει ένα πρόβλημα σχετικά με τις περιφερειακές εκτάσεις και να μην υπάρχουν εκτάσεις που προσφέρονται στον κύριο Τσόλος για να λύσει το πρόβλημά του. Θα πρέπει δηλαδή να βελτιωθεί πάρα πολύ η πρόταση διότι διαφορετικά δεν μιλάω για την πολιτική μου ομάδα αλλά για μένα προσωπικά δεν μπορεί να υπάρξει συνένεση και με μια τέτοια ανοησία δεν πρόκειται να συμφωνήσω με την γεωργική μεταρρύθμιση. Επίσης, εάν παραμείνουμε σε αυτές τις ανοησίες θα πρέπει να έχουμε δυνατότητα να διαπραγματευτούμε κατά τρόπον ώστε να υπάρξουν ε, οι ρυθμίσεις εκεί που είναι απαραίτητες και εκεί που δεν χρειάζονται ε, ε, εγώ ξέρω τι πρέπει να γίνει για να μπορέσουν να προσαρμοστούν οι εκτάσεις ε, αλλά ένας γεωργός στην Βαβαρία που προσπαθεί ήδη να εκμεταλλευτεί μία μεγάλη έκταση έχει αρκετά προβλήματα και το 7% δεν πρόκειται να το δεχθούμε επουδενή λόγο. Ευχαριστούμε Άλμπερτ. Αντιπρόεδρος ε, Σικέρσκι και μετά ο Σασαμούδη. Καταρχήν ε, ξεκινάμε από το συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται να καταλήξουμε, δεν πρόκειται να εγκρίνουμε διατάξεις που θα εφαρμοστούν πριν ε, το 2020. Ουσιαστικά φροντίζουμε από τώρα για κάποιες ρυθμίσεις που μερικές φορές δεν είναι και τόσο δίκαιες ε, και θα αφορούν τους άλλους σε μεταρρύθμιση και πράγματα που θα εφαρμοστούν μετά το 2020. Δεν κατάλαβα κύριε Καπόλο Σάντος, αυτά τα 2,5, αυτό το 2,5% είναι υποχρεωτικό από τον, πρώτο, από τον πρώτο πυλώνα για τους νέους γεωργούς. Γιατί Είπαμε αρχικά ότι η υποστήριξη προέλθει από το δεύτερο πυλώνα και μάλιστα δεν ισχύει η δεσμευτικότητα για τα κράτη-μέλη. Γιατί είπαμε δεν θέλουμε να επηρεάσουμε την ε, διακριτική τους ευχέρεια για το, ε, που θα ε, αφιερώσουν τα διάφορα κονδύλια. Γιατί έτσι είμαστε κάπως... υπαγορεύουμε στα κράτη-μέλη τι θα πρέπει να κάνουν. Και τι γίνεται με τα 100 εκτάρια γιατί νομίζω ότι είναι μεγάλη έκταση τα 100 εκτάρια. Προτιμώ τα 50 εκτάρια. Να μην φτάσουμε στα 100 εκτάρια, γιατί αν προβλέψουμε τα 100 εκτάρια, πάλι θα στρεβλώσουμε τον ανταγωνισμό. Και θα υπάρξει πάλι πρόβλημα με τις κατακαιρματισμένες γεωρικές εκμεταλλεύσεις. Επίσης το πρόγραμμα για τους ε, μικροκαλλιεργητές ή είπαμε ότι μπορούν να ενταχθούν όσοι λαμβάνουν λιγότερο από 1.500 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα κρατήσουν τις ε, τωρινές τους ενισχύσεις και ότι όλοι θα δικαιούνται τα 1.500 ευρώ. Γιατί αυτό θα επιβαρύνει πολύ τα κρατημέλη που έχουν ένα μεγάλο αριθμό μικροκαλλιεργητών. Προσοχή λοιπόν στα μέτρα που ε, θα προβλέψουμε, γιατί έτσι ίσως ε, δημιουργήσουμε και στρέβλωση ανταγωνισμού μεταξύ των Γιώργων σε ό,τι αφορά τις μεταφορές πιστώσεων μεταξύ των διαφόρων πυλώνων. Είπαμε ότι θα υπάρξει δυνατότητα μεταφοράς 10% από το πρώτο στο δεύτερο πυλώνο, ιδιαίτερα όταν ε, ε, υπάρχει, υπάρχει πρόβλημα σε χρηματοδότηση στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε αυτό το 10%. Το 5% είναι κάπως χαμηλό ποσοστό μεταφοράς. γιατί μερικές φορές επιβάλλουμε πολλές απαιτήσει και τελικά οι γεωργοί θα λαμβάνουν λιγότερα, λιγότερες ενισχύσεις από αυτές που λαμβάνουν σήμερα. Πώς θα τους το εξηγήσουμε. Επίσης είπαμε 25% για τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα από το δεύτερο πυλώνα. Είναι διαφορετικές οι διαστάσεις ε, του δεύτερου πυλώνα στις ε, διάφορες χώρες. Μερικές φορές έχουμε 38 με 48% σε ορισμένε χώρες. Σε άλλες χώρες ο δευτερο πυλωνας πυλώνας είναι 10-15% του συνολικού γεωργικού προϋπολογισμού. Οπότε ουσιαστικά θα επιβαρυνθούν οι χώρες που έχουν ε, μικρό δεύτερο πυλώνα. Θα πρέπει να εξυγχρονιστούν ταυτόχρονα και ταυτόχρονα θα πρέπει να θεωρώσουν ένα μεγάλο τμήμα του φακέλου τους για το, τα αγροπεριβαλλοντικά, κάτι που και πάλι θα τους φέρει σε δύσκολη ανταγωνιστική θέση. Θα πρέπει να κρατήσουμε μια πιο δίκαιη κατανομή. Άλλο πρόβλημα αφορά το θέμα της δημοσίευσης των πληροφοριών. Ο κόσμος, οι γεωργοί, χρειάζονται ενημέρωση πρόκειται για κρατικά δημόσια κονδύλια. Γιατί δεν θα πρέπει λοιπόν να δίνονται πληροφορίες για το ποιο δικαιούται ενισχύσει. Καλό θα είναι να δημοσιεύονται όλα αυτά τα στοιχεία, να υπάρχει διαφάνεια και να είναι προσιτές αυτές οι πληροφορίες σε όλους. Γιατί στην επιχειρηματικότητα υπάρχει τέτοιο, ε, τέτοια δυνατότητα για την ενημέρωση ότι αφορά το επίπεδο ενισχύσεων. Τώρα, για τη διαφορά μεταξύ του 3 και του 7% ε, και για το θέμα των βιοκαυσίμων, αυτό που ανέφερε ο κύριος Ντέσσε, ε, νομίζω ότι θα πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε νέους μηχανισμούς για να μπορέσουμε από το δεύτερο πυλώνα να χρησιμοποιήσουμε, να ενισχύσουμε την πρόσβαση ε, των γεωργών στις πιστώσεις. Και μάλιστα καλό θα είναι να προβλέψουμε επιδοτούμενα δάνεια από το δεύτερο πυλώνα για δυνατότητα ξυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Θα ήταν καλό να προβλέψουμε ένα τέτοιο, ένα μια τέτοια συγχρηματοδότηση κοινοτική με επιδοτούμενα δάνεια, για παράδειγμα, από το δεύτερο πυλώνα, προκειμένου η Γεωργία να εξυγχρονίσει τι εκμεταλλεύσει του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα ο Ζωζέ Μποβέ και μετά η κυρία Μαγκίνες. Τρία στοιχεία. Καταρχήν, είναι μία σκέψη σχετικά με αυτά τα οποία γίνονται στην Ουγγαρία σήμερα όπου πάνω από ένα εκατομμύρια εκτάρια ανακατανέμονται σε άτομα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη γεωργία. Πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα ε, και ε, σε σχέση με τους δραστήριους γεωργούς υπάρχει ένα πρόβλημα κατανομής των γεωργικών γεών και οι ενισχύσεις θα διανεμηθούν και στο θέμα αυτό υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχουν ολόκληρα χωριά όπου έχουν παραμεριστεί οι γεωργοί και έχουν διατεθεί οι γες σε βιομήχανους που δεν έχουν καμία σχέση. Σήμερα παρατήθηκε ο Υπουργός Γεωργίας στην Ουγγαρία σχετικά με το πρόβλημα αυτό. Υπάρχει δηλαδή πραγματικό πρόβλημα και θα δούμε πώς θα εφαρμοστούν οι ενισχύσεις. Αυτό ήταν ένα, μια υπενθύμηση απλώς επί του θέματος. Τώρα, όσον αφορά το φάκελο του κυρίου Κάπουλα Σάμπτος για το κάπινγκ και την ανακατανομή των ενισχύσεων εφόσον ε, μας, ε, έλα, ε, μας εδέχθη ο κύριος Στεφάν Λεφόλ, υπουργό Γεωργίας στη Γαλλία, ε, ε, παρουσίασε μία πρόταση η οποία πρότεινε ένα μέρος από το φάκελο του πρώτου πυλώνα 10-20% να μπορέσει να ανακατανεμηθεί για τις εκτάσεις που ήταν κάτω από τον εθνικό μέσο όρο για να υπάρχει διπλή ενίσχυση για τις μικρές εκτάσεις που είναι κάτω από τον εθνικό μέσο όρο. Ε, υπάρχει το ίδιο και σε άλλες χώρες. Μπορούμε να σκεφτούμε κάτι τέτοιο ε, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση. Δεν ξέρω πού βρίσκεστε. Εγώ ε, δεν ξέρω πού έχει φτάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ θα ήθελα όμως να ξέρω τι γίνεται. Τρίτη παρέμβαση σχετικά με το πολιτικό θέμα. Άκουσα πολύ προσεκτικά την πρόταση για το χρονοδιάγραμμα. Θα ψηφίσουμε 23-24 Ιανουαρίου στην Επιτροπή Γεωργίας και πιστεύω ότι αυτό είναι θετικό. Αντιθέτως όμως δεν νομίζω ότι είναι θετικό να ξεκινήσουμε μία συζήτηση με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν να υπάρξει η ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Όχι ότι δεν έχω εμπιστοσύνη στον εισηγητή, δεν είναι αυτό το θέμα, αλλά για πρώτη φορά θα έχουμε τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε ή στη συζήτηση ισότιμα με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα είμαστε πιο ισχυροί για να ξεκινήσουμε τη διαπραγμάτευση βασιζόμενοι σε μία ψηφοφορία στην Ολομέλεια που δεν θα είναι τελική εφόσον ξεκινά η συζήτηση αντί να ξεκινήσουμε ένα τριμερή διάλογο μεταξύ της ψηφοφορίας στην Επιτροπή Γεωργίας και της Ολομελίας. Τι θα ψηφίσουμε μετά στην Ολομέλεια, τους ε, συμβιβασμούς οι οποίοι έχουν γίνει και θα πρέπει να επανέλθουν στην Επιτροπή Γεωργίας σε σχέση με το πρώτο κείμενο που έχει υιοθετηθεί. Ε, αυτά δεν λέγονται άτυποι τριμερείς διαλογή αν υπάρχει θέση του Κοινοβουλίου θα πρέπει να υιοθετηθεί είτε μας αρέσει είτε όχι είτε υπάρξει πλειοψηφία είτε όχι αλλά πρέπει να ε, επιβεβαιώσουμε τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου είναι τα κεκτημένα μας από τη συνθήκη της Λισαβόνας και δεν πρέπει να τα απεμπολίσουμε καθοδόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ να σας χάσω αμέσως διότι, αμέσως διότι βλέπω υπάρχει σύγχυση. Εμείς θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Γεωργίας 23-24 Ιανουαρίου και φυσικά θα πάμε στην Ολομέλεια δεν πάμε το Φεβρουάριο, διότι η Ολομέλεια του Φεβρουαρίου γίνεται τι πρώτε ημέρε του Φεβρουαρίου, 6-7. Συνεπώ θα πάμε στην Ολομέλεια του Μαρτίου. Και μετά από αυτή την ψηφοφορία τη Ολομέλεια του Μαρτίου θα ξεκινήσουμε του επίσημου τριμερεί διαλόγου, παρότι υπάρχει ευρία βούληση εκ μέρου όλων και το έχουμε συζητήσει και χθε με του συντονιστέ να γίνει κάποια άτυπη συνειδρίαση, Ξεκινώντα, για παράδειγμα, από θέματα που δεν ε, ε, χαρακτηρίζονται από διχογνωμίες ε, όπως τα κείμενα εφαρμογής της Λισαβόνας. Ευχαριστούμε Ζωζέ. Ε, Μαρία Μεγκίνες τώρα και μετά Σάντρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε που μας διευκρινίσατε το χρονοδιαγράμμα, αλλά είναι σημαντικό να πούμε ότι έχουμε ελάχιστο χρόνο μετά το Μάρτιο για το επίσημο κομμάτι αυτών των συζητήσεων. Αυτό που κάνουμε τώρα λοιπόν αποτελεί το κλειδί για το αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων μέχρι τον Ιούνιο. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συζήτητες για το έργο τους. Είναι εξαιρετικά δύσκολο και γίνεται πολύ καλή συνεργασία στις ενίες ενισχύσει με τι οποίε ασχολούμαι εγώ. Δεν θα πω σε λεπτομέρειε τώρα εδώ, διότι αυτό γίνεται στις συναντήσει των σκιωδών και των πολιτικών ομάδων. Πιστεύω όμως ότι είναι σημαντικό να πούμε στους εαυτούς μας ότι αυτό δεν είναι το τελικό στάδιο της διαδικασία και ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να σκεφτεί πολύ προσεκτικά τη θέση που θα έχουμε όταν θα ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις και θέλω οι συναδέλφοι να σκεφτούν καλά αυτά τα λόγια αντί να καταλήξουν να έχουν στα χέρια τους μόνο τα τελικά συμπεράσματα της διαδικασίας να ξέρουμε τι θα βάλουμε πάνω στο τραπέζι να ξέρουμε ότι δεν θα μπορέσουμε να επιλύσουμε κάθε ζήτημα και για κάθε κράτος μέλος χρειαζόμαστε μια ευρεία προσέγγιση οι δύο δύσκολοι τομεί είναι τα μέτρα πρασινίσματος, του greening και το ζήτημα της σύγκληση, τόσο εξωτερική και εσωτερική σύγκληση. Και τα δύο αυτά ζητήματα σχετίζονται με το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Χαίρομαι λοιπόν που ψηφίζουμε τον Ιανουάριο, διότι έτσι τα πράγματα μπορεί να γίνουν λίγο... θα είναι πιο σαφή τότε από ότι σήμερα και θα θέλαμε όλοι φυσικά να συμφωνηθούν οι συμβαστικές τροπολογίες μας μέχρι τα τέλη αυτού του μήνα ή αρχές Δεκεμβρίου και για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί όσον αφορά τις εξελίξεις στο MFF. Συμπερασματικά πιστεύω ότι σημειώνουμε πρόοδο, αγχώνουμε λίγο για την κατάσταση πώς θα έχει τον επόμενο Μάρτιο και πώς θα προσπαθήσουμε να το ολοκληρώσουμε όλα αυτά μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Ακόμη και οι ίδιες οι συνεδριάσεις, η διεξαγωγή των ίδιων των συνεδριάσεων είναι δύσκολες, αλλά πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο είναι αποφασισμένο να τηρήσει αυτή την προθεσμία και να προσφέρει βεβαιότητα στους γεωργούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μαγκίνες που υπογραμμίσατε αυτή την ισχυρή βούληση του Κοινοβουλίου να επιταχύνει τις διαδικασίες όσο αυτό είναι δυνατόν για μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση. Σάντρα Γανιέτε. Και μετά κύριε Σολαϊνίτσακ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, εισηγητές μας και τους σκιώδης εισηγητές γιατί πραγματικά εργάστηκαν ε, άοκνα προκειμένου να καταλήξουμε σε συμβεστικές προτάσεις και να γεφυρώσουμε τη διάσταση απόψεων που επικρατεί μεταξύ μας για πολλά γεωργικά θέματα. Θα ήθελα να φερθώ σε ορισμένα θέματα που είναι σημαντικά για τους ε, λετονούς γεωργούς. Είναι κρίμα που δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε σαφείς συμβαστικές προτάσεις για το θέμα της σύγκλησης. Γιατί υπάρχουν πολλές προτάσεις, αλλά δυστυχώς καμία από αυτές δεν, δεν μας ικανοποιεί. Γιατί θέλουμε να ευθυγραμμίσουμε τις ενισχύσεις ε, σε χώρες που λαμβάνουν ε, κάτω από το 50% του κοινωτικού μέσου όρου. Θα πρέπει να βρούμε κάποιες ε, ειδικέ λύσεις, ώστε μετά το τέλος της μεταβατικής περίοδου οι, ε, γεωργοί μας να λαμβάνουν τουλάχιστον το 80% του κοινωτικού μέσου όρου σε αφορά τις ενισχύσεις σε ένα εκτάριο. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα εδώ στο Κοινοβούλιο μόνο, θα πρέπει να το συζητήσουμε με το Συμβούλιο ή τουλάχιστον να επιληφθεί το Συμβούλιο και να το λύσει. Άλλο σημαντικό θέμα για την Λετωνία είναι το θέμα του πρασινίσματος, όπως λέμε. Αυτή τη στιγμή το 50% του λετωνικού εδάφους ε, καλύπτεται από δάση ή από ε, οικολογικές ε, ζώνες βλάστησης μάλλον. Και μετά την ανάκτηση ανεξαρτησίας μας, ουσιαστικά χάσαμε το μισό της γεωργικής μας έκτασης. Ένα τεράστιο δηλαδή, μια τεράστια πόλια. Και μάλιστα με τις επιπλέον υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους γεωργούς, αυτοί θα υποχρεωθούν να βάλουν στην αγρανάπαυση 3, 5 έως και 7%. Δεν έχει καμία οικονομική τεκμηρίωση μια τέτοια πρόταση. Έχω υποβάλει πολλές προτάσεις και πιστεύω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα σε περιφερειακή βάση και περιπτωσιολογικά. Γιατί κάτι που είναι δυνατό στι σκανδιναβικέ χώρε ή στι βαλτικέ ε, χώρες δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί στην Ιταλία, στην ε, Ελλάδα, στι χώρε του Νότου. Και το θέμα της μεταβατικής περίοδου θα έχει ιδιαίτερη σημασία. Θα πρέπει αυτή να είναι όσο πιο βραχία γίνεται, τουλάχιστον για την Λετωνία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα της διαφάνειας, μετά το 2004 και μετά την προσχώρηση της πατρίδας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για πολλά χρόνια ακούγαμε στοιχεία για τις ενισχύσεις που δίνονται στους γεωργούς και στις ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις και όμως δεν υπάρχει σχετική απέτηση στη, από την κυρωτική νομοθεσία να δημοσιεύονται τέτοια στοιχεία, τελικά κάποια στιγμή διακόπηκαν αυτές, ε, ε, αυτές οι δημοσιεύσεις. Κάτι που δυσαρέσει τον κόσμο, γιατί πρόκειται για χρήματα των φορολογουμένων, οπότε θα πρέπει να υπάρχει ε, λογοδοσία και διαφάνεια για το πού διοχετεύονται αυτά τα κονδύλια. Επίσης δεν εξετάσαμε και τον ορισμό του ενεργού γεωργού, active farmer. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, γιατί και στην Ελετονία έχουμε ε, ενιαία, ενιαίο καθεστώς πληρωμών και σε αντίθεση με άλλες χώρες έχουμε πολλούς γεωργούς του καναπέ όπως τους λέμε, ανενεργούς πλήρως που παρόλα αυτά λαμβάνουν ενισχύσεις εφάμιλες με αυτές που λαμβάνουν και πραγματικά δραστήριοι και ενεργοί γεωργοί. Ευχαριστώ κύριο Σολέινιτσακ και μετά ο, συνα... ο Αντιπρόεδρος Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος των συζητήσεων και με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι έχουμε όλο και περισσότερες συμβαστικές προτάσεις επιτάπητος. Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνούμε ότι μας έχει μας έχουν απομείνει αρκετές εκκρεμότητες ακόμη και είναι πιο εμφανής όλο η διάσταση απόψεων και οι εντάσεις και οι που υπάρχουν μερικές φορές μεταξύ μας. Εγώ δεν είμαι και πολύ αισιόδοξο, γιατί φαίνεται ότι ενεργοποιούνται όλο και περισσότερα που εφιστούν την προσοχή μας σε πολύ σημαντικά θέματα για παράδειγμα θέματα του πρώτου πυλώνα. Εμείς ε, καταφέραμε ο πρώτος πυλώνας να συμβάλλει σε αύξηση της παραγωγής και ταυτόχρονα στην ε, προστασία του περιβάλλοντος. Αλλά τώρα, διαβάζοντας τις διάφορες συμβαστικές προτάσεις, διαπιστώνω ότι καλές είναι μεν, αλλά δεν ε, μας βοηθούν να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας και μάλιστα φαίνεται ότι περιπλέπουμε ακόμη περισσότερο την κοινή γεωρική πολιτική που γίνεται δύσκολη για τη διοίκηση ως προς τη διαχείρισή της αλλά γίνεται ε, και για τους γεωργούς και τα όρια που επιβάλλουμε και οι υποχρεώσεις που επιβάλλουμε όπως ε, επισήμανε και ο κύριος Ακέσκη δεν είναι αρκετά σαφή και συγκεκριμένα. Ε, δίνουμε τη δυνατότητα για επιπλέον επιδοτήσει στον πρώτο πυλώνα για τους νέου γεωργού αλλά το συνολικό ποσό του κάθε κράτου το περικόπτουμε. Οπότε θα υπάρξουν εντάσεις στα κράτη-μέλη. Επίσης, το ίδιο ισχύει και για τους μικροκαλλιεργητές. Σε πολλές χώρες, όπως και στην Πολωνία, δεν θα καταφέρουμε να ε, υλοποιήσουμε με επιτυχία αυτό το πρόγραμμα για τους μικροκαλλιεργητές φαίνεται ότι αυτές οι προτάσεις θα παραμείνουν στη θεωρία. Λέμε ότι θα είναι το 10% του ποσού, που σημαίνει ότι θα πρέπει διαμετρικά να περικοπεί και οριζόντια η συνολική ποσόστοση, οπότε οι περισσότεροι γεωργοί θα επιλέξουν να παραμείνουν στο ισχύον σύστημα. Φαίνεται ότι αναζητούμε συμβαστικές λύσεις που είναι ανεφάρμοστες στην πράξη. Είναι κάπως ε, ουτοπικές και θα είναι ανέφικτες για τα περισσότερα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο πυλώνα, με ιδιαίτερη ικανοποίηση διάβασα την πρόταση για τις γεωρικές ασφαλίσεις. Νομίζω ότι στον 21ο αιώνα είναι απαραίτητες τέτοιου είδους ρυθμίσεις αλλά και εκεί υπάρχουν κάποιες ε, κρεμότητες. Θα πρέπει να δούμε πώς θα συγχρηματοδοτήσουμε ή θα επιδοτήσουμε κάποια δάνεια, όπως είπε και ο κύριος Σεκέρσκι. Και οι πράσινοι, αλλά και εμείς οι σοσιαλιστές έχουμε υψηλές προσδοκίες ε, υπέρ κάποιων γεωργοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων. Στην Πολωνία έχουμε τεράστιο προϋπολογισμό για το δεύτερο πυλώνα και το 25% για τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα θα είναι ένα ποσό που θα ξεπερνάει το σύνολο του προϋπολογισμού πολλών χωρών για το δεύτερο πυλώνα. Δεν μπορούμε ad hoc να υιοθετήσουμε ένα τέτοιο μηχανισμό, γιατί υπάρχουν μεγάλες διαφορές στο εύρος του προϋπολογισμού του δεύτερου πυλώνα μεταξύ των χωρών μελών. Όλε αυτές τις διαφορές θα πρέπει να τις σταθμίσουμε. Επίσης, τα όρια για το πρασίνισμα της γεωργίας. Εκεί αναφέρονται ε, τα 10 εκτάρια, απελευθέρωση 10 εκταρίων για οικολογικούς λόγους. Καλό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά μερικοί φαίνεται φοβούνται να παραδεχτούν ότι κάτι τέτοιο σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε αν αυτό το πρόγραμμα αν θα είναι 3, 5, 7% θα εξυπηρετήσει πραγματικά το σκοπό μας. Γιατί έχουμε μια κατάσταση σήμερα ε, και πιστεύω ότι με τη νέα πρόταση θα περιπλέξουμε το διοικητικό σύστημα, θα περιπλέξουμε την υποβολή των αιτήσεων, θα έχουμε δύσκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, θα έχουμε περίπλοκο σύστημα και το ελέγχο. οπότε θέλουμε μεν πιο πράσινη, ισορροπημένη γεωργία, αλλά δεν νομίζω ότι θα καταφέρουμε το στόχο αυτό με το πρόγραμμα που προτείνεται. Για όλα αυτά τα θέματα ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε πιο διεξοδικά και πιο λεπτομεριακά και όχι μόνο ε, αφηρημένα και γενικά ή σε πολιτικό επίπεδο όπως συνηθίζουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά την ε, πρόταση του κυρίου Λαβία, είμαι σκιώδης ηγητές, ε, κάνουμε βήματα προς σωστή κατεύθυνση. Είχαμε πρόβλημα τις τελευταίες μέρες με τη δημοσίευση των προσωπικών δεδομένων των δικαιούχων. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να κρατήσουμε απόρριτα αυτά τα στοιχεία. Εγώ είμαι υπέρ της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαι δηλαδή υπέρ της δημοσίευσης των προσωπικών δεδομένων των δικαιούχων. Νομίζω ότι είναι δίκαιο κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ωραία. Ο, τώρα ο κύριος ε, Αντιπρόεδρος Βασικόφσκι και μετά ο κύριος Πόλσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι το πρόβλημά μας έγκυται στο ότι προσπαθούμε να βρούμε ένα και μόνο φάρμακο για πολλές αρρώστιες, δηλαδή μια πανάκια. Σε ό,τι αφορά τις οικολογικές ζώνες, συμφωνώ ότι ε, βλέπουμε τι γίνεται στην Γαλλία που έχουμε διαδοχή των χωραφιών, Σίτου, Αραβόσιτου. Εκεί πραγματικά υπάρχει η ανάγκη να έχουμε και πιο πράσινα οικολογικά μέρη. Το αντίθετο το έχουμε στις βαλτικές χώρες. Εκεί έχουμε πολύ περισσότερα δάση και μας λείπουν καλλιέργειες. Στην Πολωνία βλέπουμε όλο και περισσότερες οικολογικές ζώνες και όλο και πιο δυναμική ανάπτυξη, αλλά αυτό δεν με χαροποιεί ιδιαίτερα γιατί περιορίζεται η γεωργική ζώνη. Σε ό,τι αφορά τις άμεσες ενισχύσεις εκτάριο αυτό δεν εξυπηρέτησε τους ε, γεωργούς, παρόλο που έχουμε πολλές ε, οικολογικές ζώνες. Εγώ θα ήθελα, και αυτό είναι το συμπέρασμά μου από τη σημερινή συνεδρίαση, να, θα ήθελα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει κάποια στοιχεία. Ποιες αλλαγές παρατηρήσαμε μετά το 2004. Πώς ε, άλλαξαν οι αρδεύσιμες επιφάνειες στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα τέτοια στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί προβαίνουμε σε μεταρρυθμίσεις χωρίς να ξέρουμε ποια είναι η ακριβή εικόνα της παρούσας κατάστασης. Αν δεν μπορεί να τα βρει αυτά τα στοιχεία, εγώ δεν μπορώ να τα βρω αυτά τα στοιχεία, γι' αυτό ζητώ τη βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώ τροποποιήθηκε η εικόνα των αρδεύσιμων καλλιεργιών στα κράτη-μέλη τα τελευταία δέκα χρόνια. Υπήρξαν αλλαγέ, γιατί διαισθητικά... Εμ, Έχω διαπιστώσει αυτό το φαινόμενο που σας παρατήρησα, που σας εξέθεσα προηγουμένως. Το επισήμανε και η κυρία Καλινέτη. Όσο λιγότερες είναι οι άμεσες ενισχύσεις, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι οικολογικές ζώνες. Η οικολογία από μόνη της αναπτύσσεται δυναμικά, ακριβώ επειδή εγκαταλείπουν ε, τις γεωργικές εκτάσεις οι γεωργοί εξαιτία τη ανεπάρκεια των ενισχύσεων. Αλλά αυτό είναι πραγματικά επικίνδυνο φαινόμενο, γιατί αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική, θα μα λείψει το ψωμί κάποια στιγμή. Ευχαριστώ. Η Αντιπρόεδρο κυρία Πόλσον και μετά η Ελίζα Πετιέλια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τώρα θα συμμετέχω σε μια ε, συζήτηση στην οποία δεν έχω συμμετασχεί ιδιαίτερα μέχρι σήμερα για τον πυλώνα 1 αλλά θα ήθελα να αγγίξω αυτό το 7% ε, για οικολογικά αίτια. Δεν ξέρω πώς πρέπει να ερμηνεύσουμε αυτό το έγγραφο της Κομισιόν αλλά νομίζω ότι είναι προφανές ότι αυτό που συμβαίνει είναι ότι προσπαθούμε να διατηρήσουμε τη ποικιλότητα και τη γενετική κληρονομιά. Η γεωργία αφορά ουσιαστικά τη, τη θάσευση της φύσης. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε γεωργία απολύτως απελευθερωμένη από τις ιδιοτροπίες της φύσης. Είναι σπατάλη χρόνο να προσπαθούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι διαδρόμους στις αγροτικές περιοχές. Για μένα στη Σουηδία το ζήτημα αφορά περισσότερο τη δημιουργία τέτοιων διαδρόμων στη δασοκομεία, στα δάση και όχι στις γεωργικές περιοχές. Χρειαζόμαστε ε, λωρίδες γης όπου διάφορα ζώα θα έχουν τη δυνατότητα να επιβιώσουν. Διάφορα είδη και επίσης χώρους όπου μπορούμε να ε, συναντηθούμε και συγγνώμη, αλλά όπου μπορούν να συναντηθούν και αυτή είναι προϋπόθεση για να ε, διαβιβαστεί στις επόμενες γενιές το γενετικό DNA. Συνεπώς κύριε Ντες, ε, το να βάζουμε στην άκρη κάποια κομματή γης δεν ε, ικανοποιεί κάποια προϋπόθεση εδώ. Πρέπει να διατηρούμε την βιοπικιλότητα. Θα ήταν γελίο να ε, απλά να πάρουμε ένα 7% και να το βάλουμε στην άκρη. Δεν εξυπηρετεί καθόλου αυτό το σκοπό. Αυτό ήταν τώρα το, η αφετηρία μας ουσιαστικά. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι για τους περισσότερους γεωργούς το θέμα είναι να μπορέσουν να επανυπολογίσουν την αρδεύσιμη γη τους ή τη γη που έχουν στη διάθεσή τους. Αυτό το 7% είναι ε, περιθώρια ή άκρες, ε, παρυφές δασών, οτιδήποτε είναι ακτή, ε, λίμνης ή ποταμού, οχθή. Αυτές είναι οι πιο βιολογικά ενεργές Yes, αυτές πρέπει να διατηρήσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ερμηνεύσουμε ότι πρέπει να βάλουμε στην άκρη αρδεύσιμη γη εκτάσεις γεωργικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν διότι κάτι τέτοιο δεν θα εξυπηρετούσε κανέναν απολύτως βιολογικό περιβαλλοντικό σκοπό. Το ζήτημα είναι οι παρυφές, τα περιθώρια, οι άκρες, οι όχθες να είναι ε, ελεύθερες και για τους περισσότερους ενδιαφερομένους το ζήτημα εδώ είναι να επανυπολογίσουν ουσιαστικά τις εκτάσεις τους αυτό θα πρέπει να γίνει σαφές απολύτως τόσο εκ μέρους του Συμβουλίου όσο και της ε, Κομισιόν ότι το ζήτημα εδώ είναι η διατήρηση της βιοποικιλότητας σε αγροτικές περιοχές, σε γεωργικές περιοχές αυτά είναι τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν όχι απλά να μιλάμε να βάλουμε στην άκρη η γρανάπαυση Εάν ε, το ερμηνεύσουμε έτσι, τότε θα πρέπει να θέτει σε αγρανάπαυση 7% της αρδεύσης της κάθε ε, γεωργός είναι εντελώς αστείο. Είναι εντελώς εκτός πραγματικότητας. Ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε Πόλσεν, Ελίζα Μπετιέγγελ και μετά τον κύριο Γκαρσία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ καταρχήν τον εισηγητή, μάλλον τους εισηγητές και όλους τους κοιόδης εισηγητές των πολιτικών ομάδων διότι πρέπει να αναγνωρίσουμε παρόλες τις κριτικές ε, τις οποίες απευθύνουμε ότι οι συνάδελφοι αυτοί κάνουν μία δουλειά η οποία είναι αξιοπρόχτησεκτη και ε, πρέπει να βρεθούν συμβιβασμοί. Αυτό το είπαμε από την αρχή. Σχετικά με αυτά που είπε η κυρία Πάουλσεν θέλω να τα στηρίξω και να προχωρήσω και περαιτέρω. Είμαι βέβαιη ότι αν κοιτάξουμε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε κράτος μέλος έχει ένα ποσοστό δυνατοτήτων ε, διαθέσεως αυτών των οικολογικών ε, εκτάσεων και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η κοινωνία μας η οποία πληρώνει φόρους απαιτεί να υπάρχουν και οριοσμένες επιδόσεις από πλευράς των γεωργών σχετικά με το περιβάλλον και με το σχέδιο αυτό υλοποιούνται αυτές οι δυνατότητες. Το είπε η κυρία Πάουλσεν, αλλά είναι αρμοδιότης των κρατών μελών και θα χρειαστεί ίσως να ξαναυπολογιστούν, οι εκτάσεις και αυτό είναι καθήκον των κρατών μελών και ε, τέλος θέλω να παρακαλέσω όλες τις πολιτικές ομάδες όσον αφορά τα ποσοστά των οικολογικών εκτάσεων θέλω να ζητήσω να βρεθεί ένα συμβιβασμό. διότι θεωρώ ότι ένα συμβιβασμό είναι πολύ πιο σημαντικός στη διαπραγμάτευση παρά εάν βρούμε μία λύση μέσω της ψηφοφορίας και ένα συμβιβασμό εγώ προτείνω με τροπολογία το 3%, άλλοι προτείνουν πολύ υψηλότερο. Πρέπει όμως να βρούμε ένα συμβιβασμό. Ο κύριος Κάπουλα Σάμπτος μιλάει για 4-5%. Αν κάπου μπορούμε να καταλήξουμε, τότε θα έχουμε λύσει ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων και τα κράτη-μέλη θα έχουν ένα καθήκον να δουν πού βρίσκονται αυτές οι εκθέσεις. Και αυτό είναι ένα θέμα που δεν θα πρέπει πλέον να μας ε, να δημιουργεί εντάσεις. Επίσης, σχετικά με αυτό που είπε ο κύριος Κάπουλο Σάντος ή μάλλον ο κύριος ε, Ντοντάν σχετικά με την παρέμβαση και την αποθήκευση και τις επιστροφές ε, για τις εξαγωγές, τις οποίες όλοι απορρίπνουν. Νομίζω ότι εκεί υπάρχει πλειοψηφία, αλλά θα ήθελα να διατηρήσουμε τη γραμμή του προϋπολογισμού μηδενική, ώστε να υπάρχει ε, αν τη χρειαστούμε και πολύ σωστά αυτό είναι κάτι που αξίζει στους γεωργούς και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι επιστροφές για τις εξαγωγές για να διαταράξουν την αγορά αλλά μπορεί να υπάρξουν διαταραχές στις αγορές που να χρειαστούν να υπάρχει αυτή η γραμμή αυτό το κονδύλι και γι' αυτό η γραμμή του προϋπολογισμού παρακαλώ να διατηρηθεί ακόμη και μηδενική όσον αφορά τον δεύτερο πυλώνα και εδώ τα μέτρα για το περιβάλλον στη Γεωργία. Εκεί υπάρχει η μεγαλύτερη διαφορά διότι ε, υπάρχει ε, στοιχεία για το περιβάλλον στον πρώτο πυλώνα και στο δεύτερο πυλώνα για τη γεωργία και δεν θα πρέπει να αυξηθούν ήδη οι αριθμοί διότι αν κατάλαβα καλά είμαστε σε καλό δρόμο και ενδέχεται η διάκριση την οποία στην αρχή είχα κατακρίνει μεταξύ ε, βιολογικών και συμβατικών ε, επιχειρήσεων να ε, μην υπόκειται σε διακρίσεις και στη συνέχεια τα μέτρα που προβλέπονται στον πρώτο πυλώνα ο κατάλογος αυτός δεν θα ισχύσει αλλά θα υπάρξουν περιορισμένα μέτρα κατά τρόπον ώστε να είμαστε σαφείς και αν δεν υπάρχει πλέον διάκριση τότε θα μπορέσουμε να ακολουθήσουμε την οδό που προτείνει ο εισηγητής. Έχω και άλλο ένα ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν τώρα ψηφίσουμε τέλος το Μάρτιο, αν αυτό είναι εφικτό, μετά όσον αφορά το Συμβούλιο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα είμαστε ακόμη ένας ισότιμος και βαρύνων ε, συνομιλητής ή το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, θα έχουν συμφωνήσει και θα μας αγνοήσουν εάν δεν συμφωνήσουμε και προβάλλουμε τροπολογίες για τα διάφορα άρθρα. Θα ήθελα να ρωτήσω αυτό το θέμα και να ακούσω τις απόψεις αυτών που συμμετείχαν στις συζητήσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή μέχρι τώρα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για μας. Ευχαριστούμε Ελίζαμπετ. Εμείς ως Επιτροπή Γεωργίας σίγουρα θα παίξουμε το ρόλο που μας αναθέτει η Συνθήκη της Λισαβόνας. Θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε και να την άποψή μα και την ψήφο μα, ε, Κυρία Γκαρσία, Όσλινγκ και μετά έχουν εγγραφεί και άλλοι. Να προσπαθήσουμε να τηρήσουμε τους χρόνους. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Ράνς Γκαρσία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω θερμά τους ηγητές και τους σκιώδης ηγητές ε, για την αργόδη τους προσπάθεια. Η Επιτροπή μας ε, δεν έχει πλούσια εμπειρία σε μεγάλα θέματα απόφαση με το Συμβούλιο και πραγματικά το έργο ανοίγει δρόμους και είναι πρωτοπόρο από αυτή την άποψη. Όλα τα μέλη της Επιτροπής ε, Γεωργίας θέλουν ε, να δημιουργήσουν ένα πρόσφορο έδαφος για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της γεωργίας μέχρι το 2020 και από εκεί και πέρα. Θα πρέπει να δώσουμε τις βάσεις για να έχουμε μια κοινή γεωργική και κτηνοτροφική πολιτική μετά το 2020. Δεν είναι τα πρώτα 6-7 χρόνια. Θέλουμε και μετά το 2020 να έχουμε μια γνήσια και βιώσιμη ε, γεωργική πολιτική. Και αυτό το στόχο θα πρέπει να τον έχουμε κατά νου. Είναι πολύ σημαντικά τα σχόλια που ακούσαμε σήμερα. Μιλήσαμε για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει όμω ταυτόχρονα να έχουμε και μια εθνική προσέγγιση και ένα εθνικό όραμα που θα συνδυάζεται και με το κοινοτικό. Ο κύριο Καπόλα Σάντο μας μίλησε για τις μεταφορές μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα. Αναφέρθηκε σε 10-15% που θα, θα μεταφέρεται μεταξύ των πυλώνων. Η συνολική εικόνα που θα πρέπει να έχουμε θα πρέπει να ξεχνά τι εξελίξει στα κράτη-μέλη. Εγώ είμαι Ισπανίδα. Στην Ισπανία ήταν πραγματικά ταμπού το θέμα της μεταφοράς ε, μεταξύ των πυλώνων πριν από λίγα χρόνια. Ήταν απαράδεκτη οποιαδήποτε συζήτηση. Στο μεταξύ υπήρξε εξέλιξη και στην νοτροπία και μεταξύ των γεωργών. Τώρα έχουμε αλλάξει γνώμη και θεωρούμε ότι η μεταφορά κονδυλίου μεταξύ των πυλώνων είναι θετική. Βλέπετε λοιπόν ε, τι εξέλιξη υπήρξε στην Ισπανία και στην ε, εθνική προσέγγιση αλλά και στην οτροπία των γεωργών. Υπάρχουν αλλαγές και σε άλλες χώρες. Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνούμε τη γενική εικόνα και να δούμε τη διαφορά μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό το 10 ή 15% που θα επιτρέπεται να μεταφερθεί από τον πρώτο στο δεύτερο πυλώνα για αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, δεν μπορούμε να πετούμε όλα, όλο αυτό το 10% να αφιερώνεται σε αγρο, αγροπεριβαλλοντικά μέτρα. Αυτό δεν είναι ισορροπημένο, γιατί σε ορισμένε χώρε όπω την Ισπανία, ήδη πάνω από το 30% των κονδυλίων για την αγροτική ανάπτυξη αφιερώνεται σε αγροπεριβαλλοντικά μέτρα. Τώρα, αν και με τη νέα αυτή μεταφορά απαιτήσουμε τα κονδύλια να αφιερώνονται αποκλειστικά και μόνο σε αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, θα περιορίσουμε υπερβολικά τις εθνικές αποφάσεις που λαμβάνουν υπόψη και τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Γιατί σε μερικές χώρες δεν θα υλοποιηθεί αυτό το ποσό και έχει νόημα να επιβάλλουμε. Αλλά σε ορισμένε χώρε αφιερώνονται ήδη πολλά κονδύλια για τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη λοιπόν και οι τοπικέ ιδιαιτερότητε. Θα ήμουν πιο, αισιόδο, πιο ισορροπημένοι και πιο ε, γενναιόδοροι σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα των κρατών μελών να προσαρμοστούν. Α μην ξεχνούμε λοιπόν την ανάγκη ισορροπίας, γενεοδορίας και ιδιαίτερης μέρημνας ε, και προσοχής στην εφαρμογή αυτών των μέτρων. Το πιο σημαντικό πάντως είναι να εφαρμόσουμε την κοινή λογική στη μεταρρύθμιση αυτή. Γιατί αν ε, αγκιστρωθούμε σε εξτρεμιστικές ακραίες απόψεις, είτε οι πολιτικές ομάδες είτε τα κράτη-μέλη και χάσουμε την κοινή λογική θα επιδεινώσουμε την κατάσταση και τώρα αλλά και μετά το 2020 γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ενισχύσουμε τη γεωργία όχι μόνο τώρα αλλά και μετά το 2020. Ο κατάλογος του παραρτήματος ε, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είναι σαν να ε, ε, έχουμε υποβάλει ένα ευχολόγιο. Εγώ έχω μια τροπολογία για τον ε, τομέα των, ε, της ε, εκτροφής κουνελιών, για παράδειγμα. Είναι κάτι που δεν είναι σχετικά περιθωριακό, δεν ενδιαφέρει πολλές χώρες. Αλλά εκεί θα πρέπει να εφαρμόσουμε μια χειροδορία και να μην εμένουμε πεισματικά στα τοπικά ή εθνικά συμφέροντα, γιατί έτσι δεν θα προωθήσουμε την γενική μας προσπάθεια υπέρ της γεωργίας. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ισορροπημένοι, γενναιόδοροι, αυτό προσπαθώ να κάνω εγώ και ελπίζω και το ίδιο να κάνω και συνάδελφοι. τώρα. Κύριε Πρόεδρε, ενοχλήθηκα από τα λόγια του Άλμπερντε στην αρχή ενδεχομένως θεωρεί ότι πολλά από τα μέτρα είναι ανόητα. Αλλά τι θα γίνει αν κάποιος μας δηλώνει εκ προημίου ότι δεν θα συμφωνήσει στους συμβιβασμούς ε, νόμιζα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ε, ποσοστά για τις ε, εκτάσεις όπου θα υπάρχει κατά προτεραιότητα οικολογική μεταχείριση και ε, δεν είναι ο κύριος Δες ένας οποιοδήποτε, είναι ο εκπρόσωπος της μεγαλύτερης ε, πολιτικής ομάδας. Οπότε έτσι διεξάγει τις διαπραγματεύσεις για την πολιτική του ομάδα. Πώς θα καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό έτσι. Ξέρω ότι υπάρχει η Βαβαρία ένα κράτος ο κέντρο της Ευρώπης όπου όλα πάνε καλά αλλά ε, υπάρχουν και χώρες οι οποίες έχουν προβλήματα και γι' αυτό το greening πρέπει να ισχύσει να υπάρξουν οικολογικές εκτάσεις και οικολογική ποικιλομορφία και ε, δεν πρέπει να τσακωνόμαστε για το τι θα γίνει με το greening και να μην ξεκινάμε έτσι τις διαπραγματεύσεις. Τον παρακαλώ λοιπόν να το ξανασκεφτεί ε, και να ξανασκεφτεί τη θέση αυτών οι οποίοι διαπραγματεύονται συμβιβασμούς. Διότι μιλάμε ότι η ευελιξία θα μείνει στη διάκριση των κρατών μελών και θα παραμείνει greening by definition, δηλαδή μια τεράστια γραφειοκρατική δαπάνη και θα έχουμε μία σειρά κρατών που δεν θα διεξάγουν μία κοινή γεωργική πολιτική. Μπορεί ίσως να πιστεύουμε ότι όλα μπορούν να προσαρμοστούν ε, και ο καθένας να κοιτάζει ποια είναι τα μέτρα τα οποία μπορεί να ε, εφαρμοστούν στις επιχειρήσεις του. Θα πρέπει αυτό το οποίο θα συμφωνήσουμε να είναι εφικτό και εφαρμόσιμο και ε, ίσως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ε, θα πρέπει να συνδυάσουμε τα μέτρα του πρασινίσματος με τους ε, υπόλοιπους υπολογισμούς και αριθμούς. Ένα άλλο θέμα τώρα σχετικά με την υποχρέωση αναφοράς της, των πληρωμών και εδώ θα έλεγα ότι υπάρχει ούτως ή άλλως υποχρέωση διαφανείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, θα έπρεπε αυτό να εφαρμόζεται παντού. Ε, ε, δεν ξέρω αν θα το επιτύχουμε τελικά, αλλά δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Οι αριθμοί είναι αιτιολογημένοι, μπορούμε να τους ανακοινώνουμε και ε, ε γι' αυτά πληρώνουμε αυτά τα οποία δεν υπήρχαν προηγουμένως. Τέλος, ε, ευχαρίστω να ξανασυζητήσουμε το θέμα, αλλά ακούσαμε, είχαμε μία ακρόαση για το αμερικανικό γεωργικό σύστημα που έχει ένα σύστημα ασφαλίσεως και ε, προστασίας από τους κινδύνους και εάν θέλουμε να ακολουθήσουμε τέτοιες οδούς θα υπάρξει ένα συνολικό κίνδυνο για το δεύτερο πυλώνα, τον οποίο δεν μπορούμε καν να υπολογίσουμε αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορούμε ε, να στηρίζουμε τις ασφαλιστικές εταιρείες με δημόσιους πόρους. Τέλος, ε, τι είναι οι άτυπες συζητήσεις με το Συμβούλιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε. Ε, τι γίνεται άτυπα, ε, διότι δεν θέλω να γίνονται δύο φορές οι διαπραγματεύσεις, αλλά θέλω να έχουμε ορισμένους ορισμούς, διότι διαφορετικά πιστεύω ότι ορισμένοι θέλουν να μας δεσμεύσουν εκ προημίου έναντι του Συμβουλίου σε ορισμένα θέματα, και θα πρέπει όταν θα έχουμε καταλήξει σε συμβιβασμούς να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μία αξιολόγηση των επιπτώσεων των δυνατοτήτων μας. Αυτό δεν είναι δυνατόν. Ο κύριος Γκλάτενφερτερ τώρα. Ευχαριστώ. Καταρχήν ε, θα ήθελα να αναφερθώ εδώ ε, στις ποσοστώσεις ε, της Ζαχάρεως και την προσχώρηση της Κροατίας και να κάνω ορισμένα σχόλια σχετικά με την κατάσταση των εκτάσεων, γεωργικών εκτάσεων στην Ουγγαρία. Δυστυχώς δεν ε, λήφθη υπόψη ότι η Κροατία εξάγει 30.000 ε, ε, τόνους ο Ζαχάρεος και εντωμεταξύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι θα πρέπει ε, να ε, ε, εγκαταλειφθεί αυτή η παραγωγή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν περιέλαβε αυτή την ποσότητα ζαχάρεως στις διαπραγματεύσεις. Η Κροατία προσέρχεται, προσχωρεί μια σειρά ετών μετά τις διαπραγματεύσεις αυτές και αυτές οι 30.000 τόνοι δημιουργούν ένα πρόβλημα και στα κρατη και στην Κροατία διότι δεν θα υπάρχει ε, ε, πρόσβαση στην άχνη ε, ζάχαρη η οποία θα έρχεται από τη Βραζιλία και γι' αυτό θεωρούμε, θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να διατηρηθεί το σύστημα των ποσοστώσεων για τη ζάχαρη, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να ρυθμίσουμε τις 30.000 τόνους ε, εξαγωγών ζάχαρης από την Κροατία για να αποφύγουμε στρεβλώσεις του ανταλογονισμού στην αγορά για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες Ζακάρεως. Παρακαλώ αυτό να συνυπολογιστεί στην έκθεσή σας. Επίσης, θα ήθελα να σχολιάσω την κατάσταση στην Ουγγαρία. Προηγουμένως μας δόθηκαν πληροφορίες για ενδεχόμενες πολιτικές σκοπιμότητες και ελέγχθη ότι ένα εκατομμύριο εκτάρια ανακατανεμήθηκαν σε άτομα που δεν έχουν καμία σχέση με την γεωργία. Δεν είναι σωστό διότι η Ουγγαρία είναι πολύ μικρή χώρα ε, για να έχει κάποιον ο οποίος θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί ένα εκατομμύριο εκτάρια. 20.000 εκτάρια ε, κατανεμήθηκαν σε 12.000 επιχειρήσεις και οικογένειες και είδαμε ότι στο παρελθόν υπήρχαν πολύ μεγάλες ε, εκτάσεις, μεγάλα αγροκτήματα που εκμεταλλευόντουσαν δεκάδες χιλιάδων ε, εκταρίων που τώρα έχουν ανακατανεμηθεί σε μικρότερους ε, γεωργούς οι οποίοι <clears throat> είναι επιλέξιμοι μόνο εάν έχουν 50% των ε, εισοδημάτων τους ε, από την ε, γεωργία και αν μπορούν να έχουν και στο μέλλον αυτό το ποσοστό. Αυτό έγινε για να στηριχθούν οι νέοι γεωργοί και μη ένα ποσοστό αυτών των εκτάσεων εδόθη στους νέους. Θα πρέπει επίσης να αυξηθεί ε, και ε, ε, το κοπάδι για να μπορέσει ένας κτηνοτρόφος να είναι επιλέξιμος για αυτήν την κατανομή. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν επεμβάσεις κατά τον... Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Νίκολσον. Ευχαριστώ. Θα είμαι κι εγώ σύντομος, όσο μπορώ τουλάχιστον. Νομίζω ότι είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας συγκεκριμένα να δείξουν θετικό πνεύμα στο μέλλον. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να είμαστε και έντιμοι και ειλικρινείς. Γιατί με το χρονοδιάγραμμά μας που θα ψηφίσουμε εμείς τον Ιανουάριο και στην Ολομέλεια το Μάρτιο δείχνει πόσο περίπλοκη είναι η κατάσταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και κατά πάσα πιθανότητα ε, δεν θα προλάβουμε ε, μέχρι τον Ιούνιο να καταλήξουμε σε συμφωνία, παρόλο που αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που θέτουμε. Λυπάμαι που φαίνομαι ως πνεύμα διαφωνίας, αλλά δυστυχώς δεν είμαι και πολύ αισιόδοξο. Ούτε πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία για όλα τα θέματα. Ναι, που και που έχουμε συμφωνία μεταξύ ΕΛ και Σοσιαλιστών, είναι πλειοψηφία, αλλά αυτή είναι πλειοψηφία μεταξύ των δύο κομμάτων μόνο, δεν συμφωνούν οι υπόλοιποι. Όπως πολύ καλά ξέρει ο κύριος Καπόλα Σάντος, τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί αν δεν συμφωνηθούν όλα. Θα πρέπει να περιμένουμε λοιπόν τη συνολική συμφωνία. Εγώ παρακολουθώ δύο α, από τα ντοσιέ και βλέπω ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία. Και αν δεν συμπεριληφθεί το μενού του πρασινίσματος, δεν νομίζω ότι θα, θα καταλήξουμε σε οριστική συμφωνία. Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υπερψηφίσει δύο φορές αυτό το θέμα του πρασινίσματος. Θα πρέπει να τηρήσει τα συμπεφωνημένα. Άκουσα τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΕΛΚ και σίγουρα έχει το δικαίωμα της γνώμης του, αλλά και εμείς έχουμε το δικαίωμα διαφωνούμε. Είμαι από εκείνους που θεωρούμε ότι θα πρέπει να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία, να περιορίσουμε τις διοικητικές διατυπώσεις. Και από αυτά που είδα και άκουσα μέχρι στιγμής, το μόνο που θα κάνουμε ε, πιστεύω είναι ότι θα αυξήσουμε τη γραφειοκρατία, θα ενισχύσουμε τις διατυπώσεις αντί να τις μειώσουμε όπως θα θέλαμε. Και το άχθος όλων αυτών, το βάρος όλων αυτών θα τα αναλάβουν δυστυχώς θα το επομιστούν οι γεωργοί μας. Επίσης, ε, ε, ακούω αυτή την έκκληση για διαφάνεια και δημοσίευση των πάντων. Προσωπικά δεν έχω πρόβλημα. Αλλά όταν έγινε δημοσίευση στη δική μου περιοχή, μερικοί μοναχικοί και ευάλωτοι άνθρωποι υπέστησαν επιθέσεις και μάλιστα κακοποιήθηκαν από ανθρώπους που ε, διέριξαν τα σπίτια τους ε, γιατί είδαν ότι είχαν ε, λάβει κάποιες ενισχύσεις. Είμαι κι εγώ ανοιχτός στη διαφάνεια και στη δημοσίευση. Αλλά κάποιο που μένει σε 10-15 χιλιόμετρα μακριά από το αστυνομικό τμήμα, ε, ε, στο λόφο ή σε μια απομονωμένη περιοχή και μέσα στα μεσάνυχτα κάποιο διαρρήξει το σπίτι του, επικαλεστείτε απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο τη διαφάνεια. Θα πρέπει να είμαστε λογικοί λοιπόν και σε αυτό το θέμα και στα υπόλοιπα. Κοινή λογική. Έχουμε μακρύ δρόμο ακόμη να διανύσουμε, κοινό αλλά μακρύ δρόμο. Και επαναλαμβάνω και πάλι, τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί αν δεν συμφωνηθούν όλα και αυτό δυστυχώς ε, είναι κάτι που βρίσκεται σε πολύ μακρινό χρονικό ορίζοντα. Ευχαριστούμε Τζιμ, ήσουν πολύ σαφής. Άντριου τώρα και μετά Μπρίτερα μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τον εισηγητή και τους εισηγητές και να τους ευχαριστήσω για τη δουλειά τους για αυτή την πολύ σημαντική δουλειά που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Αυτές οι τεράστιες εργασίες εντάσσονται και σε ένα ανησυχητικό δημοσιονομικό πλαίσιο σήμερα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε λάβει. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Ζωζέ Μποβέ για την παρέμβασή του και για την ανακατανομή. Το ζήτημα αυτό τη σύγκληση είναι ένα ζήτημα κλειδί το οποίο συζητήθηκε. Θα μπορούσε να τροποποιήσει την παρέμβαση των μεταρρυθμίσεων στην περίοδο 14-20. Και αυτό το ζήτημα των πρώτων εκταρίων που θα μπορούσε να αλλάξει θεμελιωδώς ε, την έκταση της παρέμβασης. Όλο αυτό θα πρέπει να διευκρινίσει σωστά και με σοβαρότητα, διότι σίγουρα λαμβάνονται υπόψη κάποια από τα ζητήματα που έχουμε αναφέρει. Σίγουρα η ανάπτυξη της υπαίθρου, παρότι το ανέφερε ο Λουίς, θα ήθελα να αναφερθώ στις περιοχές φυσικών περιορισμών, με φυσικούς περιορισμούς και βάσει της πρότασης της Κομισιόν ε, για τον ορισμό τους μέσω συγκεκριμένων κριτήριων τίθενται, εξετάζονται αυτές οι περιοχές ως μεταρρυθμίσεις ή στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης. Υπάρχει το θέμα των προθεσμιών για τον ορισμό αυτών των περιοχών. Εγώ δεν είμαι υπέρ. Πιστεύω ότι πρέπει να οριστούν το συντομότερο δυνατό ώστε να ενταχθούν στι μεταρρυθμίσει. Είναι μια σημαντική πτυχή, πιστεύω, ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το ταχύτερο και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που μα προτείνεται αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα, μάλλον η πρόταση ε, για προσεύξη 50-55% των ποσοστών παρέμβασης για τα περιβαλλοντικά και κλιματικά θέματα. Πιστεύω ότι είναι καλό, αλλά θα πρέπει να το διευρύνουμε. Αυτή η προσεύξηση για τη βιολογική γεωργία, για τις ε, ζώνες Natura 2000 και τις ζώνες ε, που, στις οποίες εφαρμόζεται το πλαίσιο για τα ύδατα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει συνοχή εφόσον εφαρμοστούν μαζί. Ε, κατάλαβα καλά ότι το ζήτημα του greening ε, είναι ένα ζήτημα ε, στο οποίο έχουμε ακόμη πολύ δρόμο για συμβιβασμό. Στην παρούσα φάση πιστεύω ότι θα πρέπει να εντάξουμε και το ζήτημα της διαφοροποίησης. Αυτές οι εκμεταλλεύσεις όπου το 75%, το 75 των εκμεταλλεύσεων θα πρέπει να αποκλειστούν από το σύστημα αυτό και μετά όσον αφορά τις επιφάνειες οικολογικού ενδιαφέροντος, τις εκτάσεις οικολογικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν ισοτιμίες όσον αφορά την αξιολόγηση αυτών των εκμεταλλεύσεων και είναι σημαντικό να έχουμε ποικίλα ποσοστά ώστε να ενθαρρύνουμε όλες τις δυναμικές που σχετίζονται με συλλογικές δραστηριότητες. Αυτό έχει οικολογικό ενδιαφέρον. Προσπαθούμε σταθερά να ενθαρρύνουμε τις συλλογικές προσεγγίσεις αυτών των πτυχών. Τέλος, όσον αφορά τη διαφάνεια, υπάρχει αυτή η πρόταση Ναι, πρέπει να έχουμε διαφάνεια, αλλά θα πρέπει να παρέχουμε τα πραγματικά στοιχεία της διαφάνειας, όχι απλά νούμερα, τα οποία δεν έχουν πραγματική σχέση με κάτι. Δηλαδή, δεν έχει νόημα το κοινό, το, το ευρύ κοινό να βλέπει νούμερα χωρίς να καταλαβαίνει με τι σχετίζονται. Θα πρέπει να παρέχουμε τα πραγματικά στοιχεία ε, εκχώρησης δημοσίων κονδυλίων. Και για να ολοκληρώσω, όσον αφορά τον πρώτο πυλώνα, την κοινή οργάνωση αγορά, τα δικαιώματα φύτευσης, το ανέφερε και ο Σνταντά γρήγορα και εκεί όσον αφορά την αμπελουργία υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα και σήμερα δεν μπορούμε, τουλάχιστον ο Επίτροπος φαίνεται να έχει προχωρήσει όσον Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι ένα κομμάτι της διοίκησης θα παραμείνει πίσω και θα καθυστερεί τα αποτελέσματα της ομάδας υψηλού επίπεδου. Εκεί έχουμε ένα σημαντικό θέμα όσον αφορά την αμπελουργία, τον αμπελοεινικό τομέα. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα για το εξελίξει των επόμενων εβδομάδων δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι η διοίκηση, το τεχνικό κομμάτι θα επιβληθεί στο πολιτικό κομμάτι όσον αφορά τον αναπελλονικό τομέα. Grazie. Grazie, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε Ρίκ ε, Μπρίτε Ρέμες. Ευχαριστώ. Ήδη έχουμε ακούσει πολλά επιχειρήματα που έχουμε ανταλλάξει πολλές φορές και θα ήθελα να σας πω εδώ ότι εάν εφαρμόσουμε γεωργική πολιτική χρειάζεται για 7 χρόνια. Αυτό είναι ο χρόνος μας αλλά για τις βιομηχανίες είναι πολύ σύντομο αυτό το χρονικό διάστημα. Ε, ε, διάστημα. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται ένα κλίμα εμπιστοσύνης διότι προβαίνουν σε επενδύσεις οπότε δεν είναι δυνατόν να αλλάζουμε συνέχεια κατεύθυνση διότι αυτό πολιτικά διευκολύνει τους πολιτικούς να ευαισθητοποιούν ευνοούν τους πολίτες και εάν ε, υπάρχει μία πολιτική για μία 20 ετία και αλλάζουμε κάθε 7 ε, χρόνια την κατεύθυνση δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε πολιτική και γι' αυτό από τη μία πλευρά θέλουμε να ε, απελευθερώσουμε περισσότερο μετά λιγότερο θέλουμε περισσότερη παραγωγή με 7 χρόνια μετά θέλουμε λιγότερη παραγωγή και περισσότερη προστασία του περιβάλλοντος στις ίδιες εκτάσεις και αυτά δεν γίνονται σεβαστά στα κράτη-μέλη και ε, ε, ε, πρέπει να τους πούμε παραδείγματο χάρη να δούμε τι θα γίνει με τις αποδεσμεύσεις των πρημοδοτήσεων και πόσο θα προχωρήσουν οι διάφορες τομείς. Υπάρχουν πολλά θέματα επί των οποίων γίνονται τα ίδια και αυτό διαταράσει και την εμπιστοσύνη στην Ευρώπη και τη δουλειά μας εδώ. Πρέπει να είμαστε λοιπόν υπεύθυνοι για αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει και ε, για τους τομείς στους οποίους έχουμε επενδύσει. Όσον αφορά τη διαφάνεια, βεβαίως θέλουμε ε, οι πόροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη από φόρους να εφαρμόζονται ε, διαφανώς. Αλλά δεν θα πρέπει να βάλουμε εναντίον των πολιτών και αυτό αποδεικνύεται σαφώς από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Έχω όμως και πρόβλημα εάν προσπαθούμε να μειώσουμε τη σημασία των προβλημάτων. Πρέπει να διατηρήσουμε τους υγιείς τομείς τους οποίους έχουμε. Ε, κανείς να, πρέπει να ξέρει κανείς ε, ποια είναι η σωστή δοσολογία διότι μία ανάλατη σούπα δεν τρώγεται ούτε όμως μία πολύ αλμυρή τρώγεται πρέπει λοιπόν να διαμορφωθεί μία πολιτική η οποία θα δημιουργήσει τις σωστές κινήσεις και δεν θα πλήξει αυτά τα οποία δεν θέλουμε να πλήξουμε και ως εκ τούτου θα ήθελα να ξανασυζητήσουμε συγκεκριμένα πώς θα καταλήξουμε σε μία απόφαση η οποία θα είναι υλοποιήσιμη. Ο Herbert Dorfman και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζήτησα το λόγο μόνο διότι άκουσα τα, ε, ε, τα σχόλια του συναδέλφου Χόισλινγκ. Αντιλαμβάνουμε ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη υπάρχουν οι ε, ορισμένα ε, υπάρχουν βλάβες στο περιβάλλον τις οποίες θα πρέπει να πατάξουμε όπως στην Ιταλία, στην Ισπανία υπάρχουν περιοχές όπου ασφαλίζουμε ε, τα, ε, τις παραγωγές και οι γεωργοί πληρώνουν τεράστια ασφάλιστρα για να ασφαλίσουν τις παραγωγές τους πρέπει λοιπόν να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε και στη συνέχεια να δούμε τι περιορισμούς έχουμε σχετικά με την αντασφάλιση, ε, δηλαδή να δούμε ε, αν είναι ε, κάτι περιορισμένο εάν υπάρχουν δικαιώματα που ισχύουν σε μερικές χώρες και όχι σε άλλες και στις τελευταίες δεκαετίες απεδείχθη ε, η μία μέθοδος πιο αποτελεσματική από την άλλη όσον αφορά την ασφάλεια, η αντασφάλιση δηλαδή και οι αμοιβέ ασφαλίσεις αντί για κάποια άλλη ε, λύση. Δεν θέλουμε ε, να πλουταίνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες όταν υπάρχουν περιβαλλοντολογικές ε, ζημιές ε, και πρέπει να πούμε ότι ο τομέας αυτός δεν είναι ο πλέον προσοδοφόρος για τις ασφαλιστικές εταιρείες και πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα λύσουμε τα προβλήματα που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το τομέα. Ωραία, λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους. Ήταν πραγματικά μια πολύ σημαντική συζήτηση. Τώρα καλώ τους εισηγητές και τους και να λάβουν υπόψη όλα τα, όσα ακούσαμε σήμερα. Συχνά στις ε, γίνεται μια ε, αξιολόγηση από περιορισμένο αριθμό συμμετοχών. Εδώ είχαμε πολλούς συμμετέχοντες και πολλές απόψεις, ευρείες απόψεις και αυτό μας δίνει μια εικόνα πολύ πιο ευρεία. Προσοχή λοιπόν ε, να μην βρεθούμε στη δύσκολη θέση, να έχουμε συμβαστικές τροπολογίες που δεν θα έχουν ευρεία υποστήριξη όπως επιθυμούμε όλοι. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν αυτή η συζήτηση. Παρότι πλατιάσαμε, ευχαριστώ και την Κομισιόν που άκουσε όλους μας τους βουλευτές. Δίνω τώρα το λόγο στον Διευθυντή κύριο Πατσέκο. Ευχαριστώ. Ε, παρακαλώ σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την Επιτροπή αυτή για την εργασία σας και έχω κάποια σχόλια όσον αφορά τον κανονισμό για τις ενιαίες ενισχύσεις και την ενιαία κοινή οργάνωση της αγοράς και στη συνέχεια εφόσον συμφωνείτε αγαπητέ κύριε Πρόεδρε θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους μου για να σχολιάσουν και αυτοί τους άλλους κανονισμούς που έχουμε προτείνει. Πολύ γρήγορα. Όσον αφορά τις ε, άμεσες ενισχύσεις και το σύστημα για τους νέους εισερχόμενους, πιστεύω ότι εδώ Υπάρχει μια γενική συμφωνία για το τι πρέπει να γίνει. Ωστόσο, εμείς έχουμε έναν ενδιασμό όσον αφορά το ανώτατο όριο που θα συμπεριλαμβανόταν σε ένα τέτοιο σύστημα. Αυτό το ανώτατο όριο, αν είναι υπερβολικά υψηλό, θα μπορούσε να δημιουργήσει διακρίσεις μεταξύ γεωργών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι μια ανησυχία. Και όπως γνωρίζετε, έχουμε προτείνει ως ανώτατο όριο το μέσο Μέγεθο εκμετάλλευση, αν είναι άνω των 25 εκταρίων αλλά είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με αυτήν την Επιτροπή για την καλύτερη δυνατή λύση για το σύστημα για μικρά αγροκτήματα. Αυτό που μα απασχολεί δεν είναι να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα καταναλώνει υπερβολικά μεγάλο κομμάτι του κονδυλίου που έχουμε για τι άμεσε ενισχύσει, αλλά σίγουρα θέλουμε να έχουμε μια μέγιστη απλούστευση εδώ και ένα πλόενο εκτίμα για τους μικρούς αγρότε. Είμαστε λοιπόν στη διαθεσή σας για να συζητήσουμε και προτάσεις και για αυτό το θέμα. Τώρα, όσον αφορά το greening, το πρεσένισμα, θα έλεγα ότι συμφωνούμε με όσους είπαν ότι χρειαζόμαστε μια πιο απλή και πιο ευέλικτη προσέγγιση, αλλά κοινή, και το υπογραμμίζω, κοινή προσέγγιση είναι πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, ε, με ενθαρρύνει και η επισήμονση του κυρίου Σίγητη το να χρησιμοποιούμε ισοδύναμα αγροτικών μέτρων ως μέσα για ε, απλή και ευέλικτη προσέγγιση. Η έννοια εδώ που θεωρούμε καλή είναι ότι στα περιβαλλοντικά μέτρα γίνεται ήδη μια προσπάθεια πέραν του greening και εφόσον γίνεται κάτι τέτοιο θα μπορούμε να δούμε την επίτευξη των στόχων του greening. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα των περιοχών οικολογική εστίασης, συμφωνώ με όσους ανέφεραν ότι ο στόχος που θέλουμε να επιτύχουμε είναι η διαφύλαξη της βιοπικιλότητας. Αυτό θέλουμε να επιτύχουμε. Δεν θέλουμε να έχουμε αγρανάπαυση, θέλουμε να βρούμε μέσα ώστε συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διαφυλάσσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τη βιοπικιλότητα. Αντιλαμβανόμαστε απόλυτα ότι και η διατροφική ασφάλεια είναι ένας από τους στόχους και είμαστε έτοιμοι και έχουμε προτείνει ιδέες ε, να δούμε πώς θα μπορούσαμε να εντάξουμε τα πρακτικά μέσα επίτευξη αυτών των στόχων για παράδειγμα θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε μια συλλογική προσέγγιση αυτών των περιβαλλοντικά, ε, ε, περιεχών περιβαλλοντικών περιβαλλοντικής εστίασης, όπου ομάδες γεωργών θα επιτύχαναν συλλογικά τους ε, στόχους που έχουν τηθεί. Τέλος, κάτι που ήθελα να πω εγώ προσωπικά, από πλευρά, μου είμαστε έτοιμοι να, παρέχουμε, έτοιμοι να παρέχουμε στοιχεία για πιθανές ε, περιοχές και τις εξέλιξεις των περιοχών, την εξέλιξη των περιοχών, όπως ανέφερε ο Αντιπρόεδρος κ. Βατσόφσκι. Δίνω το λόγο τώρα στον συναδελφό μου για τσιπλέγω. Uh, Χαίρομαι που άκουσα ότι δεν υπάρχει διαφωνία σε ό,τι αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το δεύτερο πυλώνα. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέγραψε το μεγάλο αριθμό των πολύ σημαντικών τροπολογιών και του κυρίου Καπολοσάντου και των σκιωδών εισηγητών, αλλά σημειώσαμε και τα σχόλια των άλλων μελών της Επιτροπής Γεωργίας. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε κάποια θέματα για τα οποία εξακολουθεί να υφίσταται διάσταση απόψεων. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά την, ε, τη ζώνη με τα οικολογικό, οικολογικούς περιορισμούς. Έχουμε ένα σύστημα με 144 δείκτες. Ε, δεν ε, είναι εφαρμόσιμο αυτό το σύστημα. Θα πρέπει να το αλλάξουμε, αλλιώ υπάρχει τεράστιο κίνδυνος να καταβάλουμε αποζημιώσει για ζώνες που δεν υφίστανται τέτοιου φυσικούς ή άλλους περιορισμούς. Γι' αυτό αποφασίσαμε να θεσπίσουμε ένα σύστημα που θα στηρίζεται σε επιστημονικές αναλύσεις και πορίσματα και που θα λαμβάνει υπόψη βιοφυσικά κριτήρια δεν θα ήθελα να επισέλθω σε λεπτομέρειε, αλλά σα διαβεβαιώ ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία ελαστικότητα στο σύστημα. Μεταβατική περίοδο για ε, περιοχές που σταδιακά θα εγκαταλείψουν το σύστημα. Επίση, υπάρχουν κάποια άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη, όπως το fine-tuning, για να ε, εφαρμόσουν το σύστημα με βάση τις ανάγκες τους. Η περαιτέρω ε, καθυστέρηση της μεταρρύθμισης του συστήματος σίγουρα δεν είναι λύση αλλά χρειάζεται κάποια ελαστικότητα, κάποια ευελιξία για να αντιμετωπίσουμε τα ιδιαίτερα προβλήματα των κρατών μελών όπου υπάρχουν. Δεύτερο ζήτημα αφορά τη διαχείριση των κινδύνων και το δεύτερο πυλώνα. Το κατά πόσο θα πρέπει να υπάγεται στο δεύτερο πυλώνα η διαχείριση κινδύνων. Κατά τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι πολύ καλύτερο και ευκολότερο να διαχειριστούμε τους κινδύνους στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα. Ήδη σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχουν τέτοια στοιχεία συστήματος διαχείρισης των κινδύνων που προτείνεται στο δεύτερο πυλώνα με βάση την πρόταση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άλλο σημαντικό σημείο είναι ότι Εφόσον υπάρχουν στο δεύτερο πυλώνα τα μέτρα αυτά διαχείριση κινδυνών, τα κράτη-μέλη έχουν τη διακριτική ευχαίρεια να αποφασίσουν αν θα θεσπίσουν αυτό το σύστημα ή όχι. Υπάρχει μεγάλη ελαστικότητα λοιπόν και μεγάλη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών. Ενώ αν τα μέτρα του διαχείριση κινδύνων εμπίπτουν στον τρίτο πυλώνα δεν υπάρχει τέτοια ελευθερία. Μόνο με το δεύτερο πυλώνα εξασφαλίζεται αυτή η ελαστικότητα. Ε, σε ό,τι αφορά το ελάχιστο το 25% για τις ε, δαπάνες ε, που θα πρέπει να αφιερώνονται στα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα ε, με βάση το κονδύλιο της ανάπτυξης, της αγροτικής ανάπτυξης. Θα σας παραπέμπω στην αιτιολογική σκέψη 28 της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκεί αναφέρεται ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αφιερώνουν 25% τουλάχιστον των δαπανών του δεύτερου πυλώνα για τρία είδη μέτρων. Αγροπεριβαλλοντικά και μέτρα καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών, την οικολογική γεωργία και ζώνες ε, ιδιαίτερων ε, φυσικών ή άλλων περιορισμών. Η... Έγινε μια πρόταση για να καταργηθεί η πρόταση με βάση την οικονομική αναταξινόμηση, αλλά να εστιάσουμε την πρότασή μας στην ε, υλοποίηση των αποτελεσμάτων. Οπότε δεν υπάρχει τόσο ανακατανομή μεταξύ των αξώνων, αλλά δαπάνες ανάλογα με τα αποτελέσματα που επιτυχάνει ο κάθε άξονας. Σας παραπέμπω λοιπόν στην θεολογική σκέψη 28 που μιλάει για τις δαπάνες των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων. Πιστεύω ότι υπάρχει ε, η δυνατότητα, δίνεται δυνατότητα στα κράτη-μέλη ε, που μπορούν ε, να αποδείξουν τη σημασία των δαπανών και νομίζω ότι είναι και καλή η συμβαστική λύση που λαμβάνει υπόψη και τις θέσεις των μελών στο Συμβούλιο αλλά και των Ευρωβουλευτών. Ένα άλλο θέμα αφορά τη μορφή ότι δεν, υπά, δεν έχουν προβλέψει αρκετή ελαστικότητα σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των γεωργών στα διάφορα ε, συστήματα, προγράμματα και καθεστώτα. Αλλά θα ήθελα να σας υπογραμμίσω ότι ακόμη και με την ε, ισχύουσα πολιτική αγροτικής ανάπτυξης ε, του δεύτερου πυλώνα ήδη υπάρχει δυνατότητα των κρατών μελών να προσδιορίσουν κάποια χρηματοοικονομικά μέσα όπως ταμεία εγγύησης ή ταμεία δανειοδότησης. Έχουν δηλαδή ήδη τα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να θεσπίσουν μηχανισμούς και να εξασφαλίσουν συστήματα ε, για να μπορέσουν οι γεωργοί τους να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες που προβλέπουν οι προτάσεις του δεύτερου πυλώνα. Ευχαριστώ και ο λόγος στον συνάδελφο. Να κάνω μερικά σχόλια για το ζήτημα της διαφάνειας που αναφέρθηκε επίσης σε αυτή τη συζήτηση. Η Κομισιόν έκανε την πρότασή τη, θεωρώντα δεδομένο ότι η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών θέλουν διαφάνεια στι ε, γεωργικέ ενισχύσει. Επίσης έχουμε την αίσθηση ότι ο χρηματοοικονομικός κανονισμό, ο δημοσιονομικό κανονισμό που μόλις δημοσιεύτηκε καλεί τον νομοθέτη να εφαρμόσει διαφάνεια για τις γεωργικές ενισχύσεις όπως και για άλλες ενισχύσεις και επίσης θα ήθελα να αναφέρω ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν έχει απορρίψει την νομιμότητα της διαφάνειας απλά έχει επικρίνει τον τρόπο εφαρμογής της διαφάνειας στο παρελθόν. Βάσει όλων αυτών κάναμε την πρότασή μας που θεωρώ είναι ισορροπημένη και λαμβάνει υπόψη τα ζητήματα του ιδιωτικού απορρίτου. Ειδικότερα με την εισαγωγή ενός κατοφλίου που προστατεύει όσους δεν θέλουν να δημοσιοποιηθούν. Υπάρχουν ουσιαστικά έξι τύποι τροπολογιών. Πρώτον, τροπολογίες που διαγράφουν τη διαφάνεια από το νομοθέτημα, τροπολογίες που προτείνουν η διαφάνεια να εφαρμόζεται με συγκεντρωτικά νούμερα δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τέτοιες τροπολογίες, διότι θεωρούμε ότι ουσιαστικά άρουν το ζήτημα της ε, διαφάνειας και δεν αντιστοιχούν στις αρχές ε, που ανέφερα στην αρχή της ομιλίας μου. Στη συνέχεια υπάρχει η τροπολογία προτείνει ο κ. Συγητής, που ουσιαστικά σημαίνει ότι η δημοσίευση θα πρέπει να γίνεται μέσω ενός κωδικού. Και εδώ έχουμε μεγάλε αμφιβολίε κατά πόσο κάτι τέτοιο θα ήταν βιώσιμη λύση. Για ποιο λόγο, διότι η δημοσίευση με κωδικό δεν μα επιτρέπει να ασκούμε το δημόσιο έλεγχο με την ευρία έννοια των ενισχύσεων. Δεύτερον, πιστεύουμε ότι ένας κωδικός απλά θα δημιουργούσε υποψίες και περιέργεια σε όσους διαβάζουν τον κωδικό να μάθουν τι κρύβεται πίσω από τον κωδικό. Έτσι λοιπόν μπορεί να δημιουργήσουμε πολύ μεγάλη βεβαιότητα και δύσκολες συζητήσει. γιατί να μην εμφανίζουμε απλά τα ποσά, τα ονόματα και να λέμε ότι πληρώθηκε, δεν υπάρχει κανένας λόγος κάτι τέτοιο να είναι κρυφό. Θέλει το επιχείρημα, ο δημοσιονομικός κανονισμός μας ζητά να εφαρμόζουμε διαφάνεια μέσω της δημοσίευσης ονομάτων και ποσών. Δεν έχουμε λοιπόν κανένα λόγο να κάνουμε εξαίρεση. Θα θέλαμε λοιπόν να παραμένουμε πιστοί στην πρόταση που έχει γίνει. Τελευταία παρατήρηση, σε μια από τις τροπολογίες προτείνεται η δημοσίευση για διαφάνεια να γίνεται από την Κομισιόν. Εγώ θεωρώ ότι αυτό έρχεται σε αντίφαση με τον δημοσιονομικό κανονισμό που στο πλαίσιο της κοινή διαχείρισης απαιτεί από τα κράτη-μέλη να προβαίνουν σε αυτή τη δημοσίευση. Φυσικά ε, είμαστε διατεθειμένοι να βελτιώσουμε το προτινόμενο κείμενο και να συνεργαστούμε με τον εισηγητή και με οποιοδήποτε άλλο μέλος του Παρόντος Κοινοβουλίου ώστε να καταλήξουμε σε ένα καλύτερο κείμενο, μια καλύτερη λύση. Αλλά αυτά θα πρέπει κατά την άποψή μα να βασίζεται στην αρχή ότι η δημοσίευση θα γίνεται με όνομα και ποσό. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ και τους τρεις ε, διευθυντές. Έχουμε ολοκληρώσει τη συνεδρία της Επιτροπής. Ωστόσο θα ήθελα να σας παρουσιάσω να, την ε, Αντιπρόεδρο Ιζαμπελ Τιρόν που θα ήθελε να μας μιλήσει για αυτή την ιδέα της αγοράς των 27 κρατών μελών που συζητήσαμε χθε στη συνεδρία των συντονιστών. Για αυτό το λόγο λοιπόν η Επιτροπή έχει ολοκληρωθεί. Καλό την κυρία Ιζαμπελ Τουράου να παρέμβει και ταυτόχρονα σας υπενθυμίζω ότι η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα 26-27 Νοεμβρίου. Τρέχοντος ευχαριστώ.